Καλώς ορίσατε να ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε πολλοί. Ελπίζω να έχονται και οι υπόλοιποι. Uh, Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Διερμηνία, να χαιρετήσουμε και τη Σαμπίνε. Έχουμε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά, το οποίο μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε. Βεβαίω να σας υπενθυμίσω ότι μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο συνεδρίαση και να σας κάνω κάποιες σύντομες ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι θα γνωρίζετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο υπέβαλε την έκθεση για τους ε, στόχους για την εκπαίδευση, την ε, ευθυγράμμιση των προγραμμάτων, αλλά τα προβλήματα στην απόδοση. Πρόκειται για την έκθεση του 2016. Αύριο στις 29 θα γίνει παρουσίαση το πρωί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού από τον εισηγητή, τον κύριο Βόγκαν, και εμείς είχαμε ζητήσει να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε μια παρουσίαση. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε σλότ. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στους πρώτους μήνες του 2017. Θα ήθελα όμως να σας πω επίσης ότι ήδη στην έκθεση απαλλαγής για το 2015 προτείνω θα προτείνω δηλαδή και ελπίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μια τροπολογία που θα αναφέρεται και στα συμπεράσματα της έκθεσης ε, του ελεκτικού συνεδρίου προκειμένου να μπορέσουμε να επενθυμίσουμε ότι οι στόχοι της παιδείας δεν είναι μόνο ποσοτικοί, αλλά αφορούν ε, και ευρύτερες ε, παραμέτρους. Αυτό απλώς αναφορικά η Γραμματεία προσπαθεί να καθορίσει σε ποια ημερομηνία θα μπορέσει να μας γίνει παρουσίαση αυτής της έκθεσης και στη δική μας την Επιτροπή και ε, να υπενθυμίσω ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα συναντηθούμε με τον Επίτροπο Ναυράσιτς και σίγουρα θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και από αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω, θα διαβάσατε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών ε, Παιδείας και Πολιτισμού, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο πράγματα όμως, τα οποία θεωρώ σημαντικά. Εγκρίθηκε η Γενική Προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Επομένως, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον εισηγητή και την υποφαινόμενη. Και επίσης θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι ε, ζητήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού με το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή ε, Κάρτα, την e-Card των φοιτητών που θεωρήσαμε ότι πρέπει να προωθήσουμε και ε, χαιρόμαστε που έγινε επίσης και ένα αίτημα ώστε ο πολιτισμός να εμφανίζεται περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πρόγραμμα επενδύσεων ε, Juncker. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3 μετά τις ανακοινήσεις. Η, παρουσίαση της έρευνας που έγινε ε, τη ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για το βραβείο Λούξ, ε, την αποδοχή του βραβείου και τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης δεκαετίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να ευχαριστήσω στους συναδέλφους που δραστηριοποιήθηκαν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι Έχουμε την πρωτοβουλία αυτή του βραβείου Λουξ, ε, την οποία αγαπούμε ιδιαίτερα. Πρόκειται για το μόνο βραβείο που προσφέρεται από κάποιο κοινοβούλιο, ένα βραβείο κινηματογραφίας και είναι και μια ευκαιρία για να έχουμε μια πιο άμεση επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες και την κοινή γνώμη για θέματα που αφορούν τις ευαισθησίες και τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Γνωρίζετε βεβαίως επίσης ότι από το 2012 ξεκίνησαν ε, οι ημέρες ε, του βραβείου Λουξ ε, στις χώρες μέλη και μπορούμε να τις προωθήσουμε και εμείς στη χώρα μας και από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε χώρα ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτά τα τρία έργα που είναι στον, στη λίστα των φιναλίστ και, να μπορέ, και είναι μεταφρασμένα σε περισσότερες, σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος πάνω από 55 πόλεις προώθησαν τις ταινίες αυτές. Να συγχαρούμε τους τρεις φιναλίστ και το φιλμ ε, το οποίο κέρδισε, το Τόνι Edmund. Ε, ε, τους γνωρίσαμε τους σκηνοθέτε και στις συνεδριάσεις. Ήταν πάρα πολύ σημαντική βέβαια και η τελετή που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους άλλους δύο Φιναλίστε και το «Μόλις ανοίξω τα μάτια μου» και τη «Ζωή μου σαν κολοκυθάκι». Αυτή τη χρονιά είχαμε λοιπόν και πάλι μεγάλη επικοινομορφία και φαίνεται αυτό και από την ποιότητα των τριών ταινιών που ήταν στον κατάλογο των «Φιναλίστε». Η έρευνα αυτή διεξήχθη από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ. Την ευχαριστώ γιατί έχουμε παρουσία και από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ και ε, παρουσιάστηκε τις προάλλες στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση, αλλά δεν μπορέσαμε λόγω οργάνωσης του χρονοδιαγράμματος, αλλά ε, συμμετείχαμε και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήταν μαζί μου τις προάλλες εκεί. Ε, είχαμε συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού που συμμετείχαν και πρέπει να πω ότι στο τέλος αυτής της παρουσίασης ε, όπως θα γνωρίζετε, Κάποιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού εξέφρασαν κάποιε αμφιβολίε για το ίδιο το βραβείο, την οργάνωση και την προώθησή του και ε, με την ε, πρόεδρο, την κυρία Γκρέσλε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα κατ' ουσία ότι κανείς Άλλωστε, εκτός από μία πολύ μεμονωμένη ε, παρέμβαση ε, που είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι χρήσιμο το βραβείο αυτό, όλοι οι υπόλοιποι αναγνώρισαν ότι είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο, να το γνωρίσει λίγο καλύτερα η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, να προωθήσουμε περισσότερο τις ταινίε. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ε, θα προκύψουν και από την Επιτροπή Πολιτισμού που ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπου για αυτό το βραβείο. Να ευχαριστήσω τους ε, εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης ΚΟΜ. Την παρουσίαση θα την κάνει ο κύριος Αλέν Κρεσπινέ από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ, αλλά έχουμε εδώ και τον Ολιβιέ Παρνέ από το ε, ε τμήμα έρευνας του TNS που έκανε αυτή την ε, έρευνα. Αυτό που είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι ε, να ε, ρωτηθούν οι ευρωβουλευτές. Ξέρω ότι είχατε και ένα μικρό δείγμα ε, ενδιαφερομένων. Βέβαια δεν είναι εύκολο για τους βουλευτές να διαθέσουν κάποιο χρόνο για να απαντήσουν, αλλά έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό τους. Δεν ήταν όλοι βέβαια, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο απάντησε και με ποιοτικό τρόπο, δηλαδή ασχολήθηκε και με τα διάφορα σημεία. Ε, που μας προβληματίζουν. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και σας δίνω το λόγο, αλλά για την ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ που μου δίδει το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Κλάρκ δεν είναι εδώ για την άρρωση. Γι' αυτό εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης την οποία κάναμε στα πλαίσια της απαλλαγής. Μα ζητήσατε να κάνετε αυτή τη σφιγμομέτρηση ε, νόμις για να δούμε αν είναι γνωστό το βραφείο Λουξ και πώς το αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη. Και βεβαίως όλα τα ε, έγγραφα που φορούν τη μεθοδολογία είναι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Όσον αφορά την μέθοδο, η DigiCon ζήτησε από την ε, TNC Opinion να κάνει ποιοτική σφιγμομέτρηση και ποσοτική. Όσον αφορά την ποσοτική, τα 250 μέλη έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο σε διάφορες γλώσσες 137 από τα μέλη, 18% απήντησαν, πράγμα που είναι σημαντικό ως ποσοστό, εκπροσωπώντας όλα τις πολιτικές ομάδες και όλα τα κράτη-μέλη καθώς και τα δύο φύλλα. Όσον αφορά την ποιοτική σφιγμομέτρηση, σε 42 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη ε, ποσοτική ε, ανάλυση έγιναν, απεστάλησαν ερωτηματολόγια, έγιναν και διαζώσεις, ε, συνεντεύξεις σε διάφορα επίσης άτομα εκτός. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα, πρώτα απ' όλα τα ποσοτικά. Πάρα πολύ ψηλό ποσοστό γνώση του γραφείου. Ε, 98% γνωρίζουν ότι απανέμεται αυτό το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 9 στου 10 απαντούν ε, αυθόρμητοι πρόκειται για το βραβείο Λουξ. Δεύτερη διαπίστωση. Τα μέλη κατανοούν με μεγάλη σαφήνεια ποιο είναι ο τελικός στόχος. 115 πιστεύουν ότι ο στόχος είναι η πρόθεση της ε, γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας. Διευκολύνει επίσης με το ότι υπάρχει υποτιτλισμός 24 επίσημες γλώσσες ή ε, 80% όσον αφορά την ε, ε, εκτίμηση πιστεύουν ότι είναι κάτι το θετικό, διότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την πολιτιστική διπλωματία και πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν σχέσεις με τα δίκτυα ε, επικοινωνίας. Λίγοι πιστεύουν ότι είναι αρνητικό, πιστεύουν ότι δεν είναι θέμα δική του αρμοδιότητα η τέτοιου είδους βραβείων πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι ικανοποιητικό ε, σε σχέση με τους πόρους που διατίθενται ή η διαδικασία επιλογής δεν είναι σωστή. Όσον αφορά την ποιότητα, πιστεύουν οι περισσότεροι ότι το βραβείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, πολιτισμική πολιτιστικότητα και για την ε, δημιουργία δεσμών. Και βεβαίως θέλουν όλο και περισσότερα άνθρωποι να έχουν συμμετοχή. Όσον αφορά τον ε, ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Πιστεύουν ότι στα πλαίσια αυτού του κινηματογράφου το βραβείο Λουξ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο, δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες είναι ε, διαφανείς και γίνεται από σοβαρούς επαγγελματίες. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ε, ευρωπαϊκή διανομή να υποστηρίζεται και να διευκολύνεται χάρη στον υποτιτλισμό η διανομή τέτοιου είδους ταινιών. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το βραβείο Λουξ, έκαναν κάποιες υποδείξεις για τη βελτίωση της όλης διαδικασίας, θέλουν να γίνει πιο ορατό μέσω καλύτερης επικοινωνίας εντός του Κοινοβουλίου το βραβείο αυτό, θέλουν να ενθαρρυνθεί η εξωτερική επικοινωνία με καλύτερη ανημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου του κινηματογράφου και θα πρέπει να απευθύνεται σε ευρύτερο ακροατήριο υποψή και πρόεδρος όλη η διαδικασία. Επίσης, πολλοί θέλουν να υπάρχει μεταξύ των ταινιών που προτείνονται να υπάρχει μια ποικιλία που να αγγίζει περισσότερο ε, διαφορετικές ομάδες ατόμων. Αυτές ήταν οι κυρίες παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα θέλει το λόγο και ο Λιβιέ Παρνέ, ο διευθυντής ε, ε, του κέντρου που έκανε την έρευνα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα το ιδιαίτερο. Είμαι όμως στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν τη μεθοδολογία. Ωραία. Να δώσω λοιπόν το λόγο, δεν ξέρω αν θα πρώτα θέλουν το λόγο οι συντονιστές ή οι συνάδελφοι ή όποιος ζητήσει το λόγο γιατί δεν είμαστε και τόσο πολλοί. Η Σαμπίν Φερχάιεν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την μελέτη. Ήταν μια μελέτη που περιμέναμε αρκετό καιρό. Είχαν ακουστεί πολλές κριτικές για το ότι πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Θεωρώ όμως ότι η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε ανέκαθεν στην Επιτροπή Πολιτισμού το ότι δηλαδή πρόκειται για ένα βραβείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται όμως να αυξηθεί η ορατότητά του, όπως μας είπατε και εσείς για τα ποσοστά, το 8% θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό. Θεωρώ όμως ότι η μελέτη καθιστά σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία η οποία αναγνωρίζει την αξία του βραβείου Λούξ. Είναι πιστεύω ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η προώθηση της ε, πολυμορφίας, της πολυγλωσσίας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ ε, για το ότι η μελέτη αυτή μας δείχνει συγκεκριμένα στοιχεία και θα πρέπει επίσης, ε, πιστεύω, αυτό να μεταφραστεί και σε οικονομικούς όρους και σε χρηματοδότηση. Θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με όλους εσάς. Σίγουρα είναι τροφή για σκέψη αυτό. Να πω επίσης ότι η Doris Park στο παρελθόν έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει επαφές και να συσφίξει τις ε, σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και όλους τους ε, παράγοντες που συμμετέχουν έτσι ώστε να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο κοινό το βραβείο και να αναγνωριστεί η σημασία του. Ε, σίγουρα πιστεύω ότι εμείς οι ευρωβουλευτές πρέπει να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να αυξηθεί η ορατότητα του βραβείου. Είναι πολύ καλό το ότι υπάρχουν κινηματογράφοι οι οποίοι προβάλλουν αυτές τις ε, τρεις ε, ταινίες της φιναλίστ πρωτού δοθεί το βραβείο. Νομίζω πως αυτό είχε ονομαστεί Ευρωπαϊκή Κυριακή Κινηματογράφου ή μάλλον Κυριακή του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα συναδέλφων οι οποίοι θα ασχοληθούν ακριβώς με το βραβείο Λουξ, να αναλάβουν δηλαδή κάποιες πρωτοβουλίες διάδοσης του βραβείου σε χώρες οι οποίες ε, χρειάζεται να, ε, να έχει το βραβείο Λουξ μεγαλύτερη προβολή. Ελπίζω βέβαια να μην επαναληφθεί αυτή η πολύ άσχημη συζήτηση που είχαμε για το αν είναι αναγκαίο ή όχι το γραφείο Λούξ. Σας ευχαριστώ. Ναι, υπενθύμησα πριν ότι ήταν χρήσιμη συζήτηση στην Επιτροπή Κοντ, γιατί ακριβώς ε, αυτό που προέχει είναι να δούμε πώς να το προβάλλουμε και να μην το αμφισβητούμε, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Η Julie Ward. Um, I won't say much. Δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησα φέτος ότι υπήρχε ένας κινηματογράφος πολύ γνωστός στο κέντρο του Λονδίνου, ο οποίος ε, πρόβαλε τις ταινίες αυτές και πρόβαλε το βραβείο Λουξ. Ε, μέχρι πέρυσι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχε ένας ε, τοπικός κινηματογράφος στο Leeds, ο οποίος είχε δείξει τις ταινίες αυτές. Και μάλιστα επικοινώνησαν μαζί μου οι υπεύθυνοι Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει βελτίωση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίση χαίρομαι για το ότι έχει δημιουργηθεί επιτέλου και αυτή η πολιτική σύνδεση με το βραβείο Λούξ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τον κινηματογράφο ε, ως πηγή γνώσης, πηγή μάθησης. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένα project, Fred FM, το οποίο είναι ραδιοφωνικό και είναι εκπληκτικό. Είναι ένα εκπαιδευτικό ε, πρόγραμμα το οποίο προβάλλει τις ε, παλιές ε, ταινίε που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για το βραβείο Λουξ και μάλιστα τις ε, προβάλλει και έτσι ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν άτομα με αναπηρία. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν πιστεύω πω βοηθάει πάρα πολύ αυτό το project, το Fred FM αλλά και άλλα παρόμοια. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά και χρειάζεται όμω και εμεί να βρούμε περισσότερου τρόπου για να αυξηθεί η ενημέρωση του κοινού. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτό το βραβείο ω ε, πηγή μάθηση και να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο ε, τον ε, πολιτισμό. Οι εκπαιδευτικοί εδώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν για να προβάλλουν τον απολυτισμό, να συζητηθεί το θέμα, να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι αξίες της. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο γιατί έτσι θα έχουμε πολυθετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις δεν βλέπω. Θα ήθελα να πω ε, και εγώ δύο πράγματα. Καταρχάς, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω ότι σε πολλέ χώρε έγιναν προβολέ σε διάφορε πόλει, όπω έλεγε προηγουμένω και η Julie Βόρτ. Επομένως, ε, θα είναι ίσως ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και εμείς λίγο την κατάσταση, να δούμε σε ποιες χώρες γίνονται προβολές, σε ποιες δεν γίνονται, να ζητήσουμε και από τους συναδέλφους και όχι μόνο τα εθνικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πέρσι ήδη ε, είχαν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και είχαν και μεγάλη ε, προώθηση από πλευρά σα να δραστηριοποιηθούν. Ε, ορισμένες φορές βέβαια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε και τους ευρωβουλευτέ. Ε, πρέπει να πω ότι στη Ρώμη, στην πόλη μου, ε, προβλήθηκαν πολύ οι τρει ε, ταινίε ε, που είχαμε στον κατάλογο των φιναλίστε. Επίσης θα μπορούσαμε ίσω να έχουμε και κάποιες αλλαγέ στον κανονισμό. Δεν ξέρω αν συνέβη και στι δικέ σα τι πόλεις. Ορισμένε φορέ, η διανομή των τριών ταινιών Κάποιοι βέβαια εξ αυτών δεν συμφωνεί να προβληθεί η ταινία ε, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός εμπορικών ε, ε, κυκλωμάτων νωρίτερα από τις ημέρες Λουξ. πιστεύω ότι είναι σημαντικό, επιτρέψτε μου να κάνω την πρόταση, στον κανονισμό Όποιος συμμετέχει στην επιλογή Λουξ θα πρέπει να δίνει αυτή τη δυνατότητα. Καταρχάς και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη προβολή. Και κατά δεύτερον υπάρχει υποτιτλισμός σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και πιστεύω ότι και οι τρεις ταινίε θα πρέπει να κυκλοφορήσουν πολύ ε, νωρίτερα, ακόμα και αν ε, προβληθούν ε, στο σινεμά αργότερα. Υπήρξαν αρκετέ καταγγελίε επ' αυτού και επίση, κάτι άλλο θα πρέπει να διατίθεται και σε DVD. Ήταν πολύ λίγα και αρκετοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν μπορούν όλοι φυσικά να συμμετέχουν στις προβολές που κάνει το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά να μπορέσουμε να ε, ε, έχουμε και μεγαλύτερη προβολή μεταξύ των συναδέλφων. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Παντήστε να προσθέσετε, όχι. Ωραία. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι οι ταινίες είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Ε, εντάξει, μπορεί κάποιο να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο DVD. Καταλαβαίνω ότι οι διανομή ε, μπορούν να προβάλλουν αυτέ τι δικαιολογίε, ότι ορισμένε ταινίε είναι διαθέσιμε μόνο σε DVD και όχι στο κινηματογράφο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά και να ασκήσουμε κριτική σε αυτό. Αλλά νομίζω πως ε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να δει τις ταινίε αυτές και τις τρει. αν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, από τον υπολογιστή του, από το τάμπλετ, από οτιδήποτε. Δεν υπάρχει δικαιολογία δηλαδή για να μας ε, απαντήσετε ότι δεν προλάβουμε, δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Γιατί ήθελα το DVD και δεν μπορούσα να τη δω στο κινηματογράφο. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για να δει κανεί τι ταινίε αυτέ. Ναι, εντάξει, προσπαθούσα λίγο να ε, καλύψω και αυτούς που ήταν και λίγο τεμπέληδες και δεν έκανε καν αυτή την προσπάθεια. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ε, προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πολύ σημαντικό βραβείο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Μετά από αυτό λοιπόν να περάσω στο επόμενο θέμα. Το σημείο 4 της ημερησίας διάταξης την έκθεση. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η συνάδελφος Κομοντίνη. Α, συγγνώμη. Δεν σας είδα, εδώ είστε. Συγγνώμη. Η Τερές Κομοντίνη Κάρκια, η οποία είναι η συγγήτρια της γνωμοδότησης για τα μέτρα που στόχο έχουν να απο ε, τρέψουν το γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλε μορφές διάκριση των πελατών που βασίζεται σε εθνικότητα, τόπο διανομή και διαμονή, κλπ. Πρόκειται για μια πρόταση κανονισμού για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεωγραφικό αποκλεισμό και παρά το γεγονός ότι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή ΙΝΚΟ, θεωρήσαμε ότι η δική μας Επιτροπή στα στοιχεία τα οποία την απασχολούν θα πρέπει να εκφράσει την άποψή της μέσω αυτής της γνωμοδότησης. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω, δίνοντας αμέσως το λόγο στην κυρία Κομοντίνη, ότι ε, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 11 και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 24 Ιανουαρίου. Να δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω. Μάλιστα, λάβαμε λοιπόν την πρόταση κανονισμού και πιστεύω πως ο σκοπός ήταν να δούμε πώς η γλώσσα και η βιομηχανία του πολιτισμού μπορεί να τοποθετηθεί, να λάβει θέση για αυτόν τον κανονισμό και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ή να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη προστασία σε αυτή τη βιομηχανία έτσι ώστε να ανθίσει. Αυτά λοιπόν σχετικά με την πρόταση για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Καταρχάς να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να αυξήσει την πρόσβαση στα διασυνοριακά αγαθά και τις υπηρεσίες και αυτό αποτρέποντας τις έμεσες και άμεσες διακρίσεις από εμπόρους. Όταν οι διακρίσεις αυτές έχουν σχέση είτε με τον τόπο εγκατάστασης, τόπο διαμονής ε, του ε, τελικού χρήστη. Η πρόταση δεν θέλει να αποτρέψει όλες τις ε, μορφές ε, αυτής ε, της διάκρισης, αλλά μόνο εκείνες οι οποίες ε, αποτελούν ε, όπως ονομάζει, ε, αδικαιολόγητες μορφές γεωγραφικού αποκλεισμού. Η πρόταση αποκλείει τις ηλεκτρονικές δορυφορικές υπηρεσίες ε, που αφορούν κυρίως την πρόσβαση σε ε, έργα τα οποία απολαμβάνουν καθεστώς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό ήδη αποκλείεται, ήδη προστατεύονται κάποια έργα τα οποία έχουν διάφορα θέματα σχετικά με την ε, πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία έργα αυτά έχουν άμεσε επιπτώσει στον πολιτισμό και στι ε, βιομηχανίε που ασχολούνται με αυτόν. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένε εξαιρέσει ε, στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπάθησα λοιπόν να έχω γνώμονα ορισμένες προτεραιότητες και να αξιολογήσω δηλαδή πώς η Επιτροπή Πολιτισμού μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο τον κανονισμό μέσω των αρμοδιοτήτων της και στην πρώτη περίπτωση εξέτασα αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα γίνει σε δύο χρόνια από την θέση σε ισχύ και ήταν πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση θα εξετάσει και ε, το ενδεχόμενο τέτοιο περιεχόμενο που ε, προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού θα ε, συμπεριλαμβάνεται στο γεωγραφικό αποκλεισμό. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση η οποία θα ασχολείται συγκεκριμένα με τις ιδιαιτερότητες ε, των ε, θεμάτων αυτών. Πρέπει λοιπόν να το δούμε και όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, δηλαδή ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικές ε, υπηρεσίες μουσικής, πρέπει να δούμε τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν. Αυτό λοιπόν χρειάζεται λεπτομερή εξέταση έτσι ώστε να αξιολογήσουμε ε, το αν πραγματικά λαμβάνει η χώρα αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού. Τώρα, μια άλλη προτεραιότητα για εμένα, καθώς ε, εξέτασα τον κανονισμό, ήταν ο διαχωρισμός ανάμεσα στην έννοια του ε, πελάτη και του καταναλωτή, αλλά και τι βοήθεια μπορεί να απολαμβάνουν σε περίπτωση κάποιας διαφωνίας. Εδώ η Κομισιόν κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν, που αγοράζουν ε, επιγραμμικά αγαθά και υπηρεσίες, με μονομένους χρήστες, νομικά ε, πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα. Αν δηλαδή είναι ένας χρήστης, αν είναι μια εταιρεία. Στην ε, περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι startup εταιρείε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ή κάποιε άλλε εταιρικέ μορφέ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει μεμονωμένους χρήστες. Αναφέρει ότι μόνο οι μεμονωμένοι χρήστες θα απολαμβάνουν βοήθειας απέναντι στις εθνικές αρχές. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι φορείς στον χώρο του πολιτισμού είναι είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε ε, startup, είτε διάφορες ε, ενώσεις οι οποίες δεν, ε, δεν είναι νομικά πρόσωπα, θεώρησα καλύτερα να προτείνω το εξής. Αυτές οι επιχειρήσεις να λάβουν και εκείνες συνδρομή. διότι το κέρδος αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρό. Διαφορετικά, εάν συνυπολογιστούν και αυτές οι μορφές ε, ενώσεων, τότε θα, είχαν, είχε αυτό καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν θα είχαν ε, οικονομική δυνατότητα προσφυγής. Γι' αυτό λοιπόν εστιάζουμε εδώ μόνο στην εφαρμογή του κανονισμού. και όχι σε θέματα πνευματική ιδιοκτησία. Δεν θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επιλύσουμε θέματα πνευματική ιδιοκτησία, διότι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό. Αυτό που θέλουμε είναι αυτές οι ενώσεις να επωφεληθούν από τις διαδικτυακές διασυνοριακές πλατφόρμες. Το οποίο πιστεύω πως θα βοηθήσει πολύ όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού. Θα υποβάλω λοιπόν και τις σχετικές τροπολογίες, οι οποίες να σας πω πως ε, υπάρχουν για να βοηθήσουν την ε, ομαλή μετάβαση, να βοηθήσουν λοιπόν ε, τη διατύπωση του κανονισμού. Μία από αυτές αφορά το άρθρο 2 παράγραφο ε. Εδώ προτείνω να διαγραφεί ένας κατάλογος αγαθών τα οποία προτείνει η Επιτροπή. Γι' αυτό έχω προτείνει λοιπόν τη διαγραφή του καταλόγου. Έχω προτείνει τη διαγραφή διότι δεν φαίνεται πως αυτός ο κατάλογος ε, αφορά άμεσα αυτόν τον ε, κανονισμό, αυτός ο κατάλογος με τις περιπτώσεις γεωγραφικού αποκλεισμού. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς γίνεται να υπάρχει διασυνοριακή επιγραμμική πρόσβαση σε αγαθά όπως ε, το ρεύμα, το νερό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να διαγραφούν αυτά. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές σε σχέση με τις τροπολογίες. Να πω πως ε, θα χαρώ να συνεργαστώ με όλους εσάς και να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσει που κάνατε στη γνωμοδότησή σας και σα ευχαριστώ πολύ. Η Ζαμπίνε Φερχάιεν. Μία ερώτηση έχω σε σχέση με το αέριο, το ρεύμα και το νερό. Σίγουρα ε, δεν ε, έχουν άμεση σχέση με το επιγραμμικό της, ε, του κανονισμού. Όμως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα που θα μπορούσατε να μας ε, πείτε. Να, για παράδειγμα υπάρχει ένας Γερμανός ο οποίος δουλεύει στις κάτω χώρες. Έχει λογαριασμό στη Γερμανία, πρέπει να πληρωθεί από τον Ολλανδό εργοδότη του εκεί. Έχει όμως ε, έξοδα. Ποιος θα πληρώσει το ρεύμα του. Υπάρχει, υπάρχει θέμα. Ο πάροχος ο Ολλανδός θα απαιτήσει από τον Γερμανό εργαζόμενο να ανοίξει λογαριασμό στην Ολλανδία για να πληρώνει έτσι τον λογαριασμό. Ε, αυτό δηλαδή είναι ένα παράδειγμα γεωγραφικού αποκλεισμού στα συστήματα επιγραμμικών πληρωμών. Βλέπουμε λοιπόν την διασυνοριακή διάσταση του προβλήματος. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής. Και πως ε, για να ανοίξει κάποιο ε, λογαριασμό πρέπει να ε, πληρεί διάφορε προποθέσει. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα, βλέπετε. Αυτό είναι το παράδειγμα που ήθελα να σα πω. Πρώτα έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Νέκοφ. Ο κύριος Νέκοφ και μετά η Κριστίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σήμερα τα φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει να αγοράζει κανείς online. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται με τις πληρωμές που δεν ακολουθούν την ίδια τάση. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση Επιτροπής καθώς και την προσέγγιση που υιοθέτησε δεδομένου ότι υπάρχουν πρακτικές οι οποίες καταστρατηγούν την αρχή της ενιαίας αγοράς. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν βάσει της ηθαγένειας του τόπου διαμονής ή του τόπο εγκατάστασης διακρίσεις αρνητικές. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε προσκόμματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην συμπεριλάβουμε στον κανονισμό την παροχή των online ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διότι πολύ συχνά γίνεται λόγος για δημιουργίες οι οποίες προστατεύουν ε, τα πνευματικά δικαιώματα και πνευματική διοκτησία. Και όπως είπε και η συγκίτρια και συμφωνώ, τα πολιτιστικά αγαθά όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία φεριπίνα είναι ειδικά προϊόντα και θα πρέπει να κάνουμε εμπεριστατωμένη ανάλυση στον τομέα αυτό του όλου θέματος για να δούμε πώς θα ενεργήσουμε. Αναφέρεται στο άρθρο 9 ότι θα γίνει η ανηθεώρηση του κανονισμού δύο χρόνια μετά από την θέση του σε ισχύ. Και τότε θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον θα πρέπει όλα αυτά τα προϊόντα να συνεχίσουν να υπάρχουν στο ίντερνετ. Θα πρέπει φαντάζομαι να λάβουμε υπόψη και την αρχή της δευκότητας. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε, που θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε ακόμη ε, πιο δύσκολο το ε, βάρος, το άχθος, το διοικητικό για αυτές τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έτσι δημιουργούμε πρόβλημα στο διασυνοριακό εμπόριο. Υπάρχουν προβλήματα επίσης και με την αντικαταβολή κάποιων δαπανών που έγιναν με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα και η αρχή των διακρίσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα θέματα τα οποία μας ανέφερε η συγγήτρια. Εγώ θέλω να συνεργαστώ με την συγγήτρια καθώς και με τους σκιώδεις συγγητές για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Η Ελγα Τρούπερ. Ευχαριστώ Σίλβια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συγγήτρια. Γενικά θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να αντιταχθούμε στην ε, αδικαιολόγητη γεωγραφική, ε, γεωγραφικό αποκλεισμό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της ολοκληρής ενιαίας αγοράς. Έχουμε όμως εδώ ε, κάτι το οποίο είναι εντελώς αντιφατικό με αυτό το οποίο λέγεται για την ε, ενιαία εσωτερική αγορά και τον τρόπο που λειτουργεί και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πολιτιστικά αγαθά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό Συγχαίρω την Επιτροπή η οποία ανέφερε αυτό το θέμα και τόνισε το πόσο σημαντική είναι η πολιτισμική ε, πολυμορφία και τα πνευματικά δικαιώματα, την πνευματική ιδιοκτησία και ό,τι την αφορά να μην συμπεριλαμβάνεται εδώ. Ξέρουμε, παράδειγμα τους χάρη, ότι υπάρχουν ε, διάφορα ε, θέματα προχρηδανοχτοδότησης ταινιών στα πλαίσια της αρχής εδαφικότητας και των συμβάσεων που υπογράφονται. Πολύ πρόσφατα άκουσα να λέει κάποιος από την, ε, που ήταν ένας από τους ιδρυτές της Netflix που είπε ότι ναι βεβαίως μας ενδιαφέρει η πρόσβαση διασυνοριακά αλλά μόνο σε χώρες τις οποίες δεν θα πρέπει να ε, έχουμε αποκλειστικότητα την οποία θα πρέπει να την Είναι λοιπόν διαφορετική η κατάσταση ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς. όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση. Επί της αρχής λοιπόν πιστεύω ότι σωστά λέγει η Επιτροπή ότι θέλει να βελτιωθεί η κατάσταση και να μην υπάρχουν ε, ε, προβλήματα αποκλεισμού και βεβαίως θα δούμε πώς θα, δούμε, πώς θα μελετήσουμε και την αναθεωρημένη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την ιδιοκτησία. Σε αυτό όμως τον κανονισμό νομίζω ότι ε, θα πρέπει ε, αυτά τα οποία θέλει να αποκλείσει για κάποια ηλεκτρονικά μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ η κυρία Λιμπάσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω τα περισσότερα από είπε η συγκήτρια. Υποστηρίζω και την ε, τροπολογία 24 για το άρθρο 2 παράγραφος ε. Χωρίς αυτήν την ε, τροπολογία πιστεύω πως ε, περιορίζει πάρα πολύ το άρθρο. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια και θα υπερψηφίσω την τροπολογία της. Συνάδελφος Μόργανο. Ο κύριος Μόργανο, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και να πω ότι παρεμβαίνω μόνο ε, Καταρχάς για να επαναλάβω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα εδώ στην Επιτροπή. Δηλαδή, η βοήθεια από τους ε, αρμόδιους οργανισμούς ε, δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να αφορά και όλους εκείνους που μπορούν να, υποφεληθούν. Αναφέρομαι, όπως είπε και η συντάκτρια, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ε, σε νομικά πρόσωπα. μου φαίνεται ε, περίεργο να πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να υπερασπιστούν αυτούς ε, στα δικαστήρια. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια λύση λοιπόν η οποία βοηθά ε, να προστατέψουμε τους πάντες και επειδή πρόκειται και για κανονισμό πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι έχουμε εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη συντάκτηρα της γνωμοδότησης για την πολύ καλή γνωμοδότηση και τα σχόλια των ε, Ευρωβουλευτών να ξεκινήσω με το θέμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό για σας και να σας ευχαριστήσω και γιατί υποστηρίζετε την άποψή μας για ό,τι αφορά την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε ε, προστατευόμενο περιεχόμενο. Έπρεπε να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του τομέα, τους τρόπους χρηματοδότησης ε, που ορισμένε φορές βασίζεται αποκλειστικά σε αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένη βιογραφική περιοχή. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Για τη ρήτρα αναθεώρησης, την οποία ανέφερε η κυρία Μοντίνη, πράγματι πρόκειται για μια ρήτρα ανοιχτή, ε, όπως επιθυμούσατε. Ε, δεν λέμε ότι σε δύο χρόνια ή σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν αυτές οι υπηρεσίες. Είπαμε θα ε, διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό θεωρείται αιτιολογημένη και επιθυμητή η συμπερίληψή τους και από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσον είναι υποφελείς αυτές οι υπηρεσίες που είναι και ο βασικός λόγος που τις περιλάβαμε ούτως ή άλλως. Ε, εξακολουθούμε λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ το θυμίο αυτό. Όσον αφορά τις ανησυχίες σας ε, για την εφαρμογή και τους καταναλωτές σε σχέση με τους πελάτες, τον B2C και τον B2B, ε, καταρχάς Λάβαμε υπόψη τις συγκεκριμένε παρατηρήσεις που κάνετε στο θέμα αυτό και η πρότασή μας καλύπτει και το B2B και το B2C. Ε, το B2C βέβαια θέλει να καλύψει μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες ε, τείνουν να συμπεριφέρονται σαν ε, καταναλωτές διότι ο μεγαλύτερος πελάτης δεν θα πληρώσει τη συνήθη τιμή που θα καταβάλουμε εμείς αν πάμε σε μια ιστοσελίδα. Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις λοιπόν, οι οποίες σε κάποιες ε, προϋποθέσεις ε, συμπεριφέρονται ως καταναλωτές ε, και δεν θα έχουν τη συμπεριφορά μεγάλης επιχείρησης. Έχουμε αφήσει στα κράτη-μέλη σε κάποιο βαθμό τη διακριτική ευχέρεια για να εφαρμόζουν τα θέματα της επιβολής και επίσης Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε και αν εφαρμόσουν θα συνεχίσει τις υφιστάμενες δομές και εδώ έχουμε πολύ πιο καλά αναπτυγμένους μηχανισμούς για το B2C και τις σχέσεις αυτές. Είτε πρόκειται για το δίκτυο CPC που περιλαμβάνει και διασυνοριακή εφαρμογή ή τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών που προσφέρουν συμβουλές προς τις καταναλωτές. Γι' αυτό υπάρχει εδώ μια διάκριση μεταξύ καταναλωτών και πελατών, διότι για το B2B όπως γνωρίζετε υπάρχει ε, τελείως διαφορετικές δομές και θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε πάρα πολύ ε, προσεκτικά για να δούμε ε, ο, κατά πόσο θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τον κανονισμό χωρίς ε, να δημιουργήσουμε επαχθείς νέες δομές. Ε, κάποιες ε, παρατηρήσεις για τον, καθορισμό, το, για τον ορισμό των αγαθών. Ε, Αναφέρθηκε και η συντάκτρια τη γνωμοδότηση αυτό και ε, κάποιοι άλλοι, παραδείγματο χάρη για τον ηλεκτρισμό. Ε, εκεί υπήρχε κάποια σύγχυση στις συζητήσει μας με το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το πρωί ε, κατέληξαν στη γενική προσέγγιση για το σχέδιο του κανονισμού και σε εκείνες τις συζητήσεις το Συμβούλιο ε, ζητήθηκε να αφαιρεθεί η παραπομπή στο φυσικό αέριο, στο νερό και στον ηλεκτρισμό. Ο λόγο που αναφέρθηκαν είναι γιατί δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχε διατυπώσει σε άλλε κοινοτικέ πράξει για να μην υπάρχουν αποκλήσει με του ορισμού. Υπήρχε ένα ορισμό των αγαθών από την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών που χρησιμοποιήθηκε ξανά. Από τι συζητήσει, βέβαια κατέστη σαφέ ότι στα πλαίσια του γεωγραφικού αποκλεισμού δεν είναι και πολύ λογικό, διότι εδώ αναφερόμαστε στον ορισμό των αγαθών και όχι των υπηρεσιών. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ορισμός αυτός αφορά αγαθά και ε, εάν το φυσικό αέριο, το νερό και ο ηλεκτρισμός καλέπτονται ως υπηρεσίες θα πρέπει να δούμε άλλες πτυχές του κανονισμού για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Ε, στο άρθρο για παράδειγμα 4.1c μια διάταξη που θα πρέπει να οριστεί με τρόπο ώστε να τους καλύπτει ή ε, όσον αφορά τις πληρωμές, το άρθρο 5, κάποιος αναφέρθηκε σε προβλήματα πληρωμής ε, ε, αν παρέχονται υπηρεσίες σε άλλη χώρα. Βέβαια υπάρχει το πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπάρχει ο σχετικός κανονισμός και ο κανονισμός όμως αυτός για το γεωγραφικό αποκλεισμό περιέχει κάποιες προϋποθέσεις για τη μη διάκριση. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, τουλάχιστον δύο από εσά αναφέρθηκαν στην ανάγκη ε, η επιβάρηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι στο δυνατόν πιο χαμηλή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό, όπως και ε, τα κράτη-μέλη συμφωνούν. Προσπαθούμε σε όλο τον κανονισμό να διασφαλίσουμε ότι παρέχοντας ταυτόχρονα επιπλέον δυνατότητες στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες επιχειρηματίες πελάτες ε, να αγοράζουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη μικρότερη δυνατή επιβάρηση προσπαθούμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ακόμα διάκριση. Για παράδειγμα, λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ακόμα διάκριση όταν δεν υπάρχει σημαντικό επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Ευχαριστώ πολύ. Τα όσα άκουσα εδώ σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την Επιτροπή σας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη να δώσω αμέσως τον λόγο στην ε, εισηγήτρια, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να πω ότι ελπίζω και στην αναθεώρηση του κανονισμού σε δύο χρόνια θα λάβετε επαρκώς υπόψη ε, βεβαίως, γιατί είναι πολύ μικρό το, το χρονικό διάστημα, την ιδιωτερότητα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου και το γεγονότος ότι ε, πρέπει να προστατεύσουμε και τα πολιτιστικά αγαθά, και οι τροπολογίε λοιπόν που έγιναν και από τη συντάκτρια τη νομοδότηση είναι πολύ σημαντικέ ε, ω προ τα θέματα στα οποία πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο, όχι μόνο ως ε, μεμονωμένους καταναλωτέ, αλλά και πελάτε οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Και φυσικά αυτό θα σχετίζεται και με τα πνευματικά δικαιώματα και με την εφαρμογή, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και αυτά τα αγαθά. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα να κάνω για τον ε, λόγο για τον οποίο θα ήθελα να συμπεριληφθεί ο ε, πελάτης και ο καταναλωτής. Ε, δεν θέλω να υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα αγοράζουν επιγραμμικά αγαθά και υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να ε, πάνε στο δικαστήριο κάποιο, κάποια μικρή εταιρεία. Αυτό που θα ήθελα είναι οι μικρές εταιρείες, μικρές ε, ενώσεις, συνεταιρισμούς να έχουν αυτή την δυνατότητα διότι ε, λειτουργούν ως καταναλωτής. Αγοράζουν κάτι λοιπόν επιγραμμικά για δική τους χρήση όμως προσωπική, δεν το ε, πολλούν εκ νέου. Αυτό λοιπόν προτείνω στην ε, τροπολογία. Πέραν αυτού όμως ε, θα ξαναπώ ότι με μεγάλη μου χαρά θα λάβω τις προτάσεις για τροπολογίες από τους συναδέλφους και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Τροπολογίες μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, 11 η ώρα. Ψηφοφορία 24 Ιανουαρίου 2017. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε τώρα στη δημόσια κρόασή μας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Eh, sono già arrivati? Allora, Θα ήθελα να ζητήσω να έρθουν εδώ στο Προεδρείο οι τρει επιρογνώμονες. Τα ευχαριστούμε. Μαξ Βον Άμπεντροθ, εκτελεστικός διευθυντή ε, του ΕΜΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Μέσων ενημέρωση και Περιοδικών, Μάικ Χόλτερνες, δημοσιογράφος ειδικευμένος ε, στα δικαιώματα του δημιουργού, διεθνή και εθνικά, και ο Σεμπάστιαν Ντέντενς, ο, ο επικεφαλής του Uber Burda Media. Να σας καλωσορίσουμε όλους. Ε, χαίρομαι που ε, γίνεται αυτή η ακρόαση. Ελπίζω οι συνάδελφοι, ο κύριος Μαλτέζε που ζήτησε αυτή την ακρόαση να έρθει ε, το συντομότερο δυνατόν. Εμείς βεβαίως ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολύ καιρό θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Πρόκειται για μια συζήτηση για την κρίση της έντυπης δημοσιογραφίας, ε, της παραδοσιακής δημοσιογραφίας ε, στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι αυτή η ανησυχία έχει προκύψει από μια σειρά από λόγους. Προφανώς υπάρχει ε, κάτι οικονομικής φύσεως η αλυσίδα των αξιών και των ισορροπιών μεταξύ των διαφορών μέσων ενημέρωσης έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες, 20 ετία θα έλεγα εγώ, και έχει ξεκινήσει και από τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης των πωλήσεων και φυσικά υπάρχει και η ψηφιακή πρόκληση, την οποία βέβαια εκμεταλλεύτηκαν και κάποιες εφημερίδες για να μπορέσουν να διευρύνουν την ε, προσφορά ε, τους και ε, φυσικά να το πούμε και ειλικρινά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ισότιμο πεδίο ίση όρια ανταγωνισμού. Ε, η ο επαγγελματισμός ε, του δημοσιογράφου δεν γίνεται απόλυτα σεβαστούς και αυτό είναι ένα αγαθό που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφυλάξει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πολιτιστική, γλωσσική πολυμερφία, πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά πολυφωνία των μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης, όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι ένας από τους πυλώνες ε, στους οποίους εδράζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα ήθελα βεβαίω να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μια πολιτική πρόκληση. Υπάρχουν χώρες στις οποίε περιορίστηκε η ελευθεροτυπία, υπήρξαν και καταγγελίες οι οποίες έγιναν και από πλευρά Κοινοβουλίου και σε χώρε που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δεν υπάρχει και ισορροπία όσον αφορά το σεβασμό της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας ε, των ε, ε, εντύπων αλλά και των δημοσιογράφων. Και ένα τρίτο ζήτημα βεβαίως αφορά και θα θέλαμε να εξετάσουμε αυτή την κρίση και τις προοπτικές ε, οι οποίες πρέπει να ε, μπορούσαμε να, να εξετάσουμε, πώς μπορούμε να έχουμε θετικές προοπτικές για τον τύπο. Γνωρίζουμε ότι η ε, σύγχρονη σκέψη έχει προκύψει και από τις εφημερίδες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτική συζήτηση. Και αν θέλουμε ε, να είμαστε και λίγο διδακτικοί, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε ε, μία πτώση των βασικών, ε, ε, της κυκλοφορίας των βασικών εφημερίδων. Ε, η πωλήσει έχουν πέσει κατά 33%, αλλά ε, είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό για τα ε, εθνικά μέσα παρά για τα τοπικά μέσα. Ε, προφανώς οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τοπικές εφημερίδες είναι πιο συγκεκριμένες, πιο ε, ε σχετικές ε, με τα όσα γράφεται στην περιοχή του καθενός και φυσικά υπάρχει και απουσία ποιοτικών ιστοσελίδων ε, σε τοπικό επίπεδο. Ε, πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Απ' τη μια υπάρχει μια αύξηση του αναγνωστικού κοινού λόγω της ε, ψηφιακής εποχής, αλλά υπάρχει και μείωση της διαφήμισης στην έντυπη δημοσιογραφία, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρη μόνο ε, με την αύξηση που υπάρχει στην ψηφιακή διαφήμιση. Εκτιμούμε ότι η μείωση της διαφήμισης είναι περίπου στα 14 δις για 4 χρόνια, ενώ τα έσοδα στην ψηφιακή διαφήμιση είναι της τάξης των τεσσάρων δις ε, αύξησης. Επομένως, ε, οι ευρωπαϊκές εφημερίδες σίγουρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είναι πολύ δύσκολο να είναι ανταγωνιστικές και αυτή τη στιγμή δεν εγγυόμαστε και συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης και ισορροπίας. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές προκλήσεις, ε, το γνωρίζετε αυτός, για το ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν τι έχετε να μας πείτε, πώς μπορούμε να δούμε τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις προκλήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορά και τις εφημερίδες, ε, ε, το VMS, το οποίο και αυτό έχει σχέση με τα θέματα αυτά και επίσης πώς μπορούμε να εγγυηθούμε στην παρούσα κατάσταση μια πολυφωνία και ελευθερία των μέσων ε, και προστασία του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο αμέσως στον Μαξ Φον ο οποίος όπως είπαμε είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΜΑ της European Magazine Media Association που εκπροσωπεί πάνω από 15.000 εκδοτικούς οίκους σε όλη την Ευρώπη για να έχουμε μια εικόνα για την κατάσταση τη στήριξη και την ενίσχυση στον έντυπη δημοσιογραφία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και πιθανές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ε, ανέφερα προηγουμένως. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για 10 λεπτά, ο καθένας από εσάς θα έχει περίπου 10 λεπτά. Ε, θέλουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον αυτά που έχετε να μας πείτε. Παρακαλώ. Yeah, um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κώστα, για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε σήμερα για το μέλλον του ευρωπαϊκού τύπου. Στην παρουσίασή μου θα ήθελα να ασχοληθώ με τρεις ε, επιμέρους τομείς. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, μιλήσω για το περιεχόμενο ε, όχι τόσο για την, τον έντυπο, ε, τα έντυπα μέσα ή για τα ψηφιακά. Έπειτα θα ήθελα να σας μιλήσω για τις αλλαγές που διατελούνται αυτή τη στιγμή στα μέσα ενημέρωσης και τα νέα δεδομένα που έχουν εμφανιστεί στον ευρωπαϊκό τύπο, στην δυνατότητα που έχει δηλαδή να επικοινωνήσει πιο άμεσα με τους αναγνώστες και να κινητοποιηθεί σε σχέση με το περιεχόμενο. Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στον ε, νομοθέτης, το τι μπορεί να κάνει δηλαδή η νομοθεσία έτσι ώστε να εγγυηθεί ανεξάρτητο ε, τύπο, να εγγυηθεί ε, πολυμορφία και πώς δηλαδή να μην αναθέσουμε το μέλλον μας σε τρίτους, πώς δηλαδή να μην κάνουμε outsourcing. Θα δείτε λοιπόν στην παρουσίασή μου αυτήν την ανάλυση και ελπίζω κάποιες προτάσεις για λύση. Όπως ε, σας είπα και πριν, Α, μισό λεπτό. Να, νομίζω, ναι, λειτουργεί και η διαφάνεια. Όπως σας είπα, εργάζομαι για την αίμα τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Περιοδικού Τύπου, εκπροσωπούμε 15.000 εκδότες και 50.000 εκδόσεις, περιοδικές εκδόσεις. Τα μέλη μας κατά 80% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η αίμα λοιπόν προωθεί τον ελεύθερο ε, πλουραλιστικό τύπο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επίσης, είμαστε οικοδεσπότες του Future Media Lab, Ίσως το γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, ε, το διοργανώνουμε κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασχολούμαστε με το πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό που προκύπτει μετά από τις ε, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Είχαμε πριν από δέκα μέρες μία εκδήλωση σχετικά με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, θα ακολουθήσουν και άλλες και σκοπός είναι να εμβαθύνουμε σε αυτά που ε, θα ακούσετε σήμερα. Ας περάσω τώρα στο περιεχόμενο της παρουσίασής μου το οποίο αφορά τις αλλαγές που συντελούνται στο τοπίο του, των μέσων ενημέρωσης. Σε αυτό συμμετέχει ενεργά και ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής είναι αυτός που αλλάζει. Όχι μόνο όμως ο καταναλωτής, αλλά και αλλάζει η τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στον έντυπο τύπο και στο διαδικτυακό και στα κινητά τηλέφωνα ότι ε, έχουν γίνει πάρα πολλέ αλλαγέ και ότι κυρίως τα έντυπα μέσα είναι συμπληρωματικά μαζί με τα ψηφιακά. Βλέπετε εδώ τον ε, κύκλο ενός 24ωρου, ε, ενός ε, χρήστη. Ο χρήστης θέλει να έχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο σε ενημέρωση, σε μέσα και βλέπετε πως οι επιλογές του είναι ένα σύνολο από έντυπα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε καταναλωτής έχει συγκεκριμένη προσωπική χρήση και πιστεύουμε ότι αυτός που θα πιάσει το σφιγμό του καταναλωτή θα είναι αυτός που θα επιτύχει στον ε, κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Τώρα, από επιχειρηματικής άποψης μπορούμε να δούμε το πώς ε, λειτουργούν ε, συμπληρωματικά τα έντυπα μέσα και τα ψηφιακά. Βλέπουμε σε σχέση με τις συνδρομές και τις πωλήσει, αλλά και τις διαφημίσεις ότι, είναι, ότι κατανέμεται 50-50 το μερίδιο. Στα ψηφιακά μέσα τώρα πάνω από το 95% των εσόδων προέρχονται από διαφημίσεις και ε, το, τα, τα έσοδα κατά κεφαλήν στα ψηφιακά μέσα είναι πολύ μικρότερα από εκείνα των έντυπων μέσων. Χρειάζεται δηλαδή ε, να υπάρχουν 8 ψηφιακοί χρήστες για να, ε, για να καταναλώσουν αυτό που καταναλώνει ένας μόνο χρήστης έντυπων μέσων ενημέρωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά έντυπου και ψηφιακού τύπου. Τώρα, στα περιοδικά, στο περιοδικό τύπο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει αύξηση κυκλοφορίας περιοδικών, ιδιαίτερα ε, για συγκεκριμένα θέματα, εξειδικευμένος περιοδικός τύπος. Αυτό βλέπουμε ότι κρατά μείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία πληθώρα περιοδικού τύπου που ε, αφορά διάφορους ε, τομείς, ενημέρωση, εξειδικευμένα θέματα, business to business. Περνάμε τώρα στο τοπίο του ανταγωνισμού. Από τη μία, ο παράγοντας επιτυχίας για μια επιχείρηση στην Ευρώπη είναι το τι κάνεις δηλαδή για να τραβήξεις αναγνώστες. Πώς καταφέρνεις να παραμείνεις σχετικός, να παραμείνεις επίκαιρο και να προσελκύσεις ε, τους αναγνώστες αλλά και να τους κρατήσεις. Και επίσης πώς μπορείς να μεταφράσεις το αναγνωστικό σου κοινό σε χρήμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυξανόμενος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο και να σας εξηγήσω κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχάς, πώς θα προσελκύσεις αναγνώστες. Ε, Αυτή την εποχή είναι σχεδόν αδύνατον να εξυπηρετείς αποκλειστικά ε, μία κοινότητα αναγνωστών, όπως γινόταν κάποτε με τα έντυπα μέσα βλέπουμε ότι οι αναγνώστες ε, έχουν τελείως προσωπικές προτιμήσεις και προσωπική χρήση των ε, μέσων ενημέρωσης. Επιλέγουν οι ίδιοι το πότε και το πού και το πώς θα ενημερωθούν. Υπάρχουν ε, λοιπόν διάφορες πλατφόρμες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν αυτές τις επιθυμίες των αναγνωστών. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί έχουν τη δυνατότητα να ε, έχουν συνεχή πρόσβαση στον αναγνώστη. Και αυτή είναι μια απειλή που ε, αντιμετωπίζει ε, ο έντυπος τύπος. Μετά, υπάρχει και η δυνατότητα της χρηματικής αποτίμησης του περιεχομένου. Δηλαδή, Υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν μετάφρασης των αναγνωστών, του αναγνωστικού κοινού σε χρήμα, σε οικονομικά ωφέλη και αυτό δημιουργεί διάφορες διαταραχές στο αναγνωστικό κοινό. Εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε σαφέστατα ποιο είναι το πρόβλημα. Πάνω από 70% της, αγοραστική, της, της αξίας που δημιουργούν οι εκδότες πηγαίνει σε φορείς εκτός ε, του κλάδου των ε, μέσων ενημέρωσης. Μιλάμε για ε, διαφημίσεις, μιλάμε για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Google, Facebook, Twitter κτλ. Εκείνοι εξαργυρώνουν λοιπόν ε, τα ωφέλη μέσω των διαφημίσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι φορείς σε αυτόν τον χρόνο και με τα ωφέλη που μπορείτε να δείτε. βρίσκεται λοιπόν ο ευρωπαϊκός τύπος. Εδώ θα ήθελα να δω μαζί με σας τον πιθανό αντίκτυπο στα, στον, ε, στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Εάν παραμείνουν όσο έχουν τα πράγματα, το αναγνωστικό κοινό θα περάσει στις ε, κοινωνικές πλατφόρμες για την ενημέρωσή του. Αυτή η τάση θα αυξηθεί. Βέβαια, τα πράγματα δεν μένουν στάσιμα και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να σας ε, ενημερώσω γι' αυτό. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε ε, όπως είμαστε τώρα, τότε θα δούμε αυτή την αύξηση. Ποιες είναι οι συνέπειες. Και για τους εκδότες έντυπων μέσων ε, θα είναι δυσκολότερο να προσελκύσουν και να συγκρατήσουν αναγνώστες. Θα ε, περάσουν σε τομείς που δεν μπορούν να ελέγξουν και επίσης θα δυσκολευτούν να ε, έχουν έσοδα από τις ε, εκδόσεις τους. Αυτές λοιπόν είναι οι συνέπειες ως προς το περιεχόμενο και ως προς το έγκυρο περιεχόμενο και ως προς την ε, διάθεση ανεξάρτητης, αμερόληπτης πληροφορίας για τον αναγνώστη. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως, ας είμαστε επικοδομητικοί. Φυσικά πρέπει να δράσουμε. Υπάρχει αυτή η ανάγκη για δράση από διάφορους φορείς και από τις ε, εταιρείες μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ήδη προσπαθούν εδώ και κάποια χρόνια με σχετική επιτυχία να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, είτε μέσω της συνεργασίας. Συνεργασία όχι μόνο μεταξύ εκδοτών, αλλά και ε, ανάμεσα σε εκδότες και πλατφόρμες διάδοσης, όπως το Google, το Facebook κτλ. Σίγουρα χρειάζεται ε, περισσότερη δουλειά, όμως έχει γίνει η αρχή. Πρέπει να καταφέρουν λοιπόν αυτήν την οικονομική αξία να την ε, προσελκύσουν. Τώρα, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή της ε, χρηματοδότησης. Θεωρώ πως ε, είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση εδώ. Όμως, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες των εκδοτών, γιατί το νομοθετικό πλαίσιο είναι επίσης περιοριστικό. Εδώ εσείς έχετε τη δυνατότητα να διευκολύνετε την, ε, τον ίσο ανταγωνισμό, να διευκολύνετε την ε, διασφάλιση πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης ε, της Ευρώπης, έτσι ώστε τα έντυπα μέσα να μπορέσουν να επιβιώσουν και η ενημέρωση να μην ανατεθεί σε τρίτους, εκτός Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν από νομοθετική άποψη τι όπλα έχουμε στη φαρέτρα μας, Έχουμε την οδηγία για το οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε με τις προτάσεις για το φόρο προστιθέμενης αξίας και την οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Η οδηγία αυτή επηρεάζει τον τύπο με τις διάφορες νέες προτάσεις που έχουν εισαχθεί έτσι ώστε να ε, διασφαλιστεί πως τα διαφημιστικά έσοδα θα διατίθενται σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς για να διασφαλίσουμε τον πλουραλισμό. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί για την... Ε, ραδιοτηλεόραση ιδιαίτερα και εδώ σε αυτό το γράφημα μπορείτε να δείτε ότι η τηλεόραση τα τελευταία 8 χρόνια ε, παρουσιάζει αυξημένα έξοδα, πολύ περισσότερα από τα έσοδα του, ε, των έντυπων μέσων, τα οποία αντιθέτως έχουν μειωθεί εξαιτία αυτού που σα περιέγραψα πιο πριν, την έλλει τη έλλειψη χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται δράση σχετικά με αυτό. Μετά, Υπάρχει η οδηγία σχετικά με την ε, προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι για εμάς θα ήταν μία δυνατότητα ε, opt-out στα διάφορα cookies που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες ενημέρωσης στο Google, το Facebook ε, για τον υπολογιστή του χρήστη, το καλύτερο. Αυτές λοιπόν οι πλατφόρμες ε, χρησιμοποιούν αυτά τα cookies έτσι ώστε να ε, αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να τον παρακολουθούν. Χρειάζεται λοιπόν η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον να διασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία των δεδομένων αυτών τι βρίσκεται τώρα υποσυζήτηση ε, και τι προβλέπει η οδηγία για την ε, ιδιωτικότητα. Προβλέπεται λοιπόν ένα συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο όμως μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Εάν αλλάξουμε τελείως και πάμε σε ένα καθεστώς opt-in, αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν οι πόρτες για τις ε, μικρές ε, εταιρείε ε, με ΜΜΕ, οι οποίες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτό το σύστημα Δεν θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν αυτή, την οποία έχουν μεγαλύτερες εταιρείε με μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Δεν θα γίνουν λοιπόν ελκυστικές για τον αναγνώστη. Τέλος, θα ήθελα να περάσουμε τα δύο τελευταία θέματα, φόρο προστιθέμενης αξίας. Ε, περιμένουμε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα για να μειώσει το ΦΠΑ στον τύπο, στις εταιρείες ε, τύπου. Υπάρχει στήριξη από εσάς και θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη αυτή. Από όσο γνωρίζουμε θα δρομολογηθεί αυτό η οδηγία και θα, προσπαθεί, θα γίνει μια προσπάθεια να μεταφραστούν σε ε, οικονομικά έσοδα, ε, τα διαφημιστικά έσοδα σε αυτές τις πλατφόρμες. Ο συνάδελφος τώρα θα, συνεχίσει πάνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα εγώ κλείνοντας να σας ε, ευχαριστήσω για την στήριξη που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα και να σας ζητήσω να συνεχίσετε να μας στηρίζετε και στον κανονισμό για το ΦΠΑ και στις οδηγίες για τα οπτικοακουστικά μέσα και το φορό προστιθέμενης αξίας. Χρειάζεται αυτή η στήριξη έτσι ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν μια, μιας δημοκρατικής κοινωνίας και πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Ε, και, και εγώ και οι συνάδελφοι έχουμε πολλά πράγματα να σας ρωτήσουμε. Ε, φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλές παρεμβάσεις. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Μάικ Χόλτενες, ε, δημοσιογράφο ειδικευμένο σε δικαιώματα του δημιουργού σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, θα ήθελα να κάνω έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό σε μια αντιπροσωπεία από ένα σχολείο, σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Ε, το σχολείο από το οποίο έρχονται αυτά τα παιδιά είναι ε, το ε, σχολείο στο Αματρίτσε. Ξέρετε ότι το Αματρίτσε είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μαλτέζε, ο οποίος είχε την πολύ ωραία ιδέα να προσκαλέσει εδώ στις Βρυξέλλες για να γνωρίσουν από κοντά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαθητές και σπουδαστές ε, από μια περιοχή που ε, πλήγει. Ε, χαίρομαι που η κυβέρνησή μας φρόντισε αμέσω να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν το σχολείο τους και πάλι στο Αματρίτσε. Πρόκειται για παιδιά που είναι από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και το Λύκειο Ελπίζω λοιπόν να είναι πολύ καλή αυτό για το μέλλον. Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Πρώτα ε, παρασχέθηκαν κάποια λιόμενα, τώρα ε, ελπίζουμε να ξεκινήσει το χτίσιμο του νέου σχολείου. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας σταθούμε. Εγώ έχω πάει ήδη στο Ματρίτσε, πήγαν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά θα επιστρέψω. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. E Ευχαριστώ και τώρα να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μάικ Χόλτερνες, είπαμε δημοσιογράφος, ε, σας εξήγησα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Επειδή ξεκίνησα κάποια στιγμή να γράφω τα σχόλιά μου, ε, πρέπει να πω ότι το 2016 ε, ε, με οδήγησε σε σχόλια τα οποία αντανακλούν την κοινωνία και την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον ίσως ε, για κάποιους από εσά να σας πω δύο λόγια για τον εργασιακό βίο ενός δημοσιογράφου ελεύθερου επαγγελματία. Μέχρι πρόσφατα έγραφα ε, μια χιουμεριστική στήλη σε ένα ε, περιοδικό για τις επιστήμες ε, μια περιγραφή που δεν άρεσε καθόλου στο κοινοβούλιο στο Westminster όταν του συστήθηκα. Την Τετάρτη συνήθως έδινα το άρθρο μου και μετά έπεφτα για ύπνο την Πέμπτη επειδή ήμουν freelance ε, πήγαινα στο γραφείο για να αντικαταστήσω τον, ε, τον συντάκτη της στήλη που έλειπε σε διακοπές. Άνοιγα, ε, ανοίγω λοιπόν το Εμίλιο και ξαφνικά κάποιο έλεγε ποιο το έγραψε αυτό. Και επομένω το ξανάγραφα όλο από την αρχή και άρχισα να ελέγχω όλα τα στοιχεία και την ορθογραφία. Μετά το έδινα σε έναν δεύτερο συντάκτη, sub editor του λέμε στην Αγγλία, ο οποίος έκανε ένα δεύτερο έλεγχο. Ε, ξανά έγραφε πράγματα, πράγματα που και εγώ και ο συντάκτη μου είχαμε διορθώσει και μετά σκεφτόμουν θυμόμαστε τον ταλέπορο τον αναγνώστη που δεν ήξερε ε, όλο αυτό το ιστορικό και απλώ θα τη διάβαζε και θα πίστευε ότι είναι ψευδή. Ε, και μετά αυτό θα το έστερνε και πάλι στον ε, αρθρογράφο, ο οποίο θα ε, διόρθωνε κάποιε απλοποιήσει και θα τα έστελνε σε έναν άλλο συντάκτη, ο οποίο θα το έλεγε ένα άλλο συντάκτη Και όλα αυτά για μια χιουμοριστική στήλη. Και ε, αυτό ε, σας δείχνει πάρα πολύ σημαντικό, ε, πόσο σημαντική είναι η έντυπη δημοσιογραφία τα άρθρα, όπως και να φτάνουν ε, στους ε, ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η δημοσιογραφία είναι σημαντική. Η βασική θεωρία της δημοκρατίας είναι ότι εξαρτάται, ε, επαφείται στους πολίτες, να έχουν πρόσβαση δηλαδή οι πολίτες σε σωστή ενημέρωση και τελειώς πώς θα ψηφίζουν λογικά. Ε, βέβαια, ε, κάποιοι δεν ψηφίζουν παρόλη την έντυπη ε, δημοσιογραφία που υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν άρθρα, να υπάρχει αρθρογραφία. Κάτι το οποίο ε, να ε, είναι γραπτό, γιατί ε, μισή ώρα ενημέρωση στην τηλεόραση είναι λιγότερο από 3.000 λέξεις, ούτε καν ένα άρθρο λοιπόν δεν είναι. Και χρειαζόμαστε και στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να βασίζουν οι πολίτε στι αποφάσεις τους και τις ζωή τους, στις πολιτικές του αποφάσεις. Χρειάζονται κάτι μεγαλύτερο και δεν μπορούν να επιβιώσουν με 140 χαρακτήρε του Twitter το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ε, ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαδικτύες συνεργασίες οι οποίες βγάζουν μια περιουσία ε, πουλώντας διαφημίσεις δίπλα στο δημιουργικό έργο ανθρώπων και ε, αυτό γίνεται εις βάρες τους. Και δύο από αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αρκετά στην Ευρώπη και είναι ένα δίπολο. δεν είναι μονοπόλιο, είναι αυτόν τον δύο το μονοπόλιο και ε, όλο ένα και περισσότερο επισημαίνεται το πρόβλημα της συγκέντρωσης της εξουσίας σε ένα ή δύο ε, μέσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δυο μεσα και πλευρά πρέπει να πω ότι χρησιμοποιείται από το ε, management για να μειώσουν τις ε, ε, τους ανθρώπους που απασχολούν και τους μισθούς που τους δίνουν και σε πολλές περιπτώσεις ε, χρησιμοποιείται και ως ε, εφαρμογή του πολιτικού ε, θέλω του ιδιοκτήτη κάθε φορά. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική σχέση σε αυτό το χάρτη τον οποίο είχα την προηγούμενη εβδομάδα από την σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας. Αυτός είναι ο χάρτης λοιπόν που μας δείχνει ε, τα διάφορα μέσα και ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες προς τα μέσα ενημέρωσης και ε, την ισχύ των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων. Τη δυνατότητα δηλαδή οι γράφοντες να προστατεύουν αυτά που γράφουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπάρχει κάποια ε, προστασία. Η Γερμανία και η Φιλανδία έχουν από τους ισχυρότερους ε, και έχει πολύ μεγαλύτερη την εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι το κείμενο είναι ένα έργο τέχνης. Αλλά στην πρακτική εφαρμογή λείπουν πολλά, όπως ε, μας λένε οι συνάδελφοι από την Ελλάδα. Και ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ότι ο βασικός κανόνας τον οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου είναι ότι όταν διαβάζουμε τουλάχιστον κάποιες βρετανικές εφημερίδες, την Daily Mail, την Daily Telegraph πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι οι πρώτες τρεις παράγραφοι ε, είναι ουσιαστικά η άποψη του συντάκτη και μετά ξεκινούν τα νέα. Έτσι γίνεται συνήθως η αρχή της συνταξίας, αυτά τα έντυπα. το 1990 όταν μόλις είχε εμφανιστεί το διαδίκτυο και το είχα διαβάσει όλο γιατί 9 σελίδες ήταν όλες και όλες μας είχαν υποσχεθεί ότι το διαδίκτυο θα οδηγήσει στη χρυσή εποχή της δημοκρατίας. Άμεση επικοινωνία, πολίτης με πολίτη θα επικοινωνεί, θα υπάρχουν δημοψηφίσματα για τα πάντα. Θα πατάμε ένα κουμπί και θα ψηφίσουμε για, ό,τι θέλουμε. Η υπόσχεση αυτή αποδείχθηκε φρούδες ελπίδες, ε, πολλές ε, ε, ψευδείς ειδήσει, πολλές προκαταλήψεις. Ε, το 1986 ε, απέκτησα την πρώτη μου ε, σύνδεση στο διαδίκτυο. Ήταν κάτι πριν από το, τη διαδικτυακή επικοινωνία. Είχαμε την CompuPress τότε και τότε εγώ εργαζόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είπα γιατί υπάρχει προστασία της ελευθεροτυπίας στην πρώτη τροπολογία. Ήταν, το είπα αυτό 9 το βράδυ, 8 η ώρα το πρωί είχα 4, 4 δοκίμενα, 4.000 λέξεων που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει προστασία. Και ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για την ε, εμπορική και, ε, ε, διαφήμιση και πώς πρέπει να προστατεύονται αυτά. Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος πραγματικά αποτελεί πρόκληση και νομίζω ότι επήγει να γίνει αυτή η συζήτηση. Κάποιοι ε, τηρούν αυτή την υπόσχεση, κάποιοι την παραβίασαν, κάποιοι κερδίζουν, αλλά το να είναι διαθέσιμα τα πάντα χωρίς καμία πληρωμή ε, θα οδηγήσει υποτίθεται στη χρυσή εποχή της ελεύθερης ενημέρωσης. Ε, η απάντηση μου είναι βέβαια ότι η ελεύθερη ενημέρωση αξίζει κάθε σεντ που πληρώνεται γι' αυτό. Και θα μπορούσατε να κάνετε το εξή πείρασμα απόψε. Μπορείτε να αναρτήσετε μια σελίδα στη Wikipedia και να ορίσετε την, έννοια, την anti anti-social media. Μέσα σε μερικά λεπτά θα εμφανιστεί κάποιος και θα σας πει ότι δεν έχετε παραθέσει πηγές. Ε, η Wikipedia υποτίθεται ότι είναι αυτό το μεγάλο εργαστήριο στο οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να δώσει το χρόνο του ελεύθερα και να ενημερώνει όλους ελεύθερα. Και τελικά εξαρτάται απόλυτα από το έργο επαγγελματιών ε, ε, συγγραφέων. Τίποτα δεν παραμένει στην ιστοσελίδα εκτός και αν παραπέμπει στο έργο κάποιου όπως εγώ για παράδειγμα. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πολύ δύσκολη να την απαντήσει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει. Χρειαζόμαστε επαγγελματίε δημοσιογράφου, ανθρώπου που αφοσιώνονται, που αποκτούν εμπειρίε, που προσπαθούν και έχουν την εμπειρία να φιλτράρουν τα σκουπίδια και να ε, κρατήσουν τη σημαντική πληροφορία και ε, θα φροντίσουν να αποκτήσουν αυτέ τι δεξιότητε. Ιδίω στον αγγλόφωνο κόσμο, οι συνάδελφοί μου ε, ε, και χρόνια με κορόιδευαν. Μία από τις αγαπημένες μου στιγμές ήταν όταν αναφερθήκα στο φιλόσοφο Μπλούνο Λατόρ και τον έφερα στο ε, γραφείο ενός μικρού εβδομαδιαίου ε, περιοδικού και ε, μου είπε «Α, εδώ κατασκευάζετε την αντικειμενικότητα, θα μπορούσα να παρατηρήσω όταν τη φτιάχνετε». Δεκάδε άνθρωποι ξαφνικά δεν μπορούσαν να το σκεφτούν. Τρία άνθρωποι που είχαν σκεφτεί τι είναι αλήθεια και έγραφαν, ε, έπιασαν το κεφάλι του με τα χέρια του και συνέχισαν ε, να προσπαθήσουν να διορθώνουν τις ε, εκθέσεις, τις, τα κείμενα που είχαν. Η αλήθεια υποτίθεται ότι είναι η πραγματική ε, ομορφιά, είπε ο Καντ, και προσπαθούμε ακόμα να το κρατήσουμε αυτό. Και τώρα ξαφνικά μπορεί κάποιο να μα πει ότι Α, μαμά δεν μ' αρέσει ή είναι ψέματα όλα αυτά. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι αρνούνται ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή και δεν διαβάζουν οτιδήποτε ε, διαφωνεί με την άποψή τους η δημοσιογραφία προσπαθεί να είναι ε, κάτι το οποίο θα τα διορθώσει αυτά. Βέβαια είναι η πρώτη προσέγγιση του προσχεδίου της ιστορίας, αλλά κάνουμε τουλάχιστον μια προσπάθεια. Και η διαδικασία της αρχισυνταξίας που σας ανέφερα προηγουμένως μας δείχνει αυτό που οι φιλόσοφοι θα αποκαλούσαν μια ε, προσέγγιση συνέπειας. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να ε, επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτού του οποίου πιστεύουμε και να το τεκμηριώσουμε έννοια του δημοσιογράφου ρεπόρτερ είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει κάποιος, ο οποίος, ε, να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα δίνει ένα άρθρο, θα το ελέγχει κάποιος και θα αποφασίζει κάποιος ότι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Όχι κάτι το οποίο θα πουλήσει ένα εξαιρετικό διαφημιστικό ένθετο, αλλά θα προσθέσει κάτι το οποίο χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες. Ανέφερα προηγουμένως ότι ε, οι διοικήσεις των έντυπων προσπάθησαν ε, να ε, αναλάβουν οι δημοσιογράφοι το κόστος ε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ε, δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε τοπικά έντοπα πολύ δύσκολα μπορούν ε, να ε, βρεθούν στο δικαστήριο γιατί δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν. Λειτουργούν χωρίς εποπτεία διότι σημαίνει ότι έγιναν πάρα πολλές περικοπές λόγω της κρίσης και τα λεφτά που παίρνουν είναι γελία. Επομένως, από την άλλη υπήρχε και το θέμα της επιβολής συμβολέων για τους δημοσιογράφους. Ε, υπάρχει ένα έντυπο με το οποίο συνεργαζόμουν και έλεγε ότι πρέπει να ε, απαρνηθώ οποιοδήποτε δικαίωμα ότι κάποιο άρθρο ήταν δικό μου είτε το έγραψα εγώ και να θεωρείται ιδιοκτησία της εφημερίδας. Πώς θα βγάλω εγώ λεφτά μα δεν ξέρουν ότι το τάδε άρθρο ήταν δικό μου. Αυτό ξεκίνησε το 1995 με τη δική μου εμπειρία με ένα ε, περιοδικό για υπολογιστέ που ήθελε να ε, υπογράψω οτιδήποτε θα, ότι οτιδήποτε θα έγραφα δεν είναι δική μου πνευματική ιδιοκτησία. Ε, βέβαια υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητε και στι Ηνωμένε Πολιτείε και στο Ιρλανδικό Δίκαιο. Κάποιοι εκδότε ε, τους οποίους γνωρίζω προσπαθούν να κάνουν διάφορα τα οποία του παρέχει η εθνική του νομοθεσία. Τώρα, δεοντολογικά. Ε, το να μπορούμε να αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι σωστό και από δεοντολογική σκοπιά εξαρτάται από την οικονομική εξασφάλιση που έχουν οι δημοσιογράφοι. Εάν για παράδειγμα είχα απάντηση για το τι ακριβώς θα κάνουμε, ε, εγώ θα ήμουν πιο πλούσιος από το Google. Θα σας δώσω ε, κάτι το οποίο είναι φήμη. Ε, υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος προσεκλήθη από την Google για να συζητήσει για την εξαιρετική τεχνολογία και του δόθηκε εντύπωση ότι δεν τους ενδιαφέρουν πια τα χρήματα. Προσπαθούν απλώς να διαμορφώσουν τον κόσμο γιατί έχουν αρκετά χρήματα. Το σχέδιο κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία υποτίθεται ότι ζητά δικαιώματα ε, γειτονίας για τους εκδότες ε, των εφημερίων. Ξέρετε τις λεπτομέρειες φαντάζομαι ε, το Google, οτιδήποτε χρησιμοποιεί θα πρέπει να το πληρώνει. Φαντάζομαι θα το αναφέρει περαιτέρω συνάδελφο συνάδελφος στη συνέχεια σας έχουν φαντάζομαι βομβαρδίσει με ισχυρισμούς ότι αυτό είναι εις βάρος του διαδικτύου και δεν σας επιτρέπει να μπείτε εσείς από το blog του Κοινοβουλίου και να δείτε μια πηγή. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, είναι ψευδοπρόβλημα αυτό και ε, είναι η παρανοϊκή ανάγνωση της πιο ε, ε, άσχημης δικαστικής διαμάχης που θα μπορούσε να προκύψει από αυτή την υπόθεση. Τι συμβαίνει τώρα, η Google ενδιαφέρεται αρκετά και ε, τόσο που ε, βγήκε στο προσκήνιο. Ε, πριν από χρόνια ήμουνα σε μια συνεδρίαση στο Westminster και ρώτησα ποιος εκπροσωπεί την Google και κάποιοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα πλέον όμως κάνει ε, lobbying απευθείας η Google και συνάντησα αρκετούς λομπίστες που κάνουν παρουσιάσεις στη Γερμανία. Και μάλιστα σε κάποια περίπτωση ήταν περήφανοι που πέρασε η νομοθεσία στη Γερμανία που, ε, που έλεγε ότι πρέπει να δέχονται ε, περιεχόμενο και ε, επομένως είναι πλέον άδεια και είπανε σε εφημερίδες δώστε μας την άδεια για μηδενικό ποσό γιατί αλλιώς θα χάσετε τους αναγνώστες σας γιατί δεν θα σας βάζουμε εμείς στις πρώτες σελίδες και δεν θα σας βρίσκουν. Οι Ισπανοί νομοθέτες ε, αποφάσισαν ότι ε, θα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πληρωμή αντί να υπάρχει υποχρεωτική άδεια. Και αν πάτε στο news.google.is θα δείτε μία ανακοίνωση από την Google που λέει ότι δεν υπάρχει πια Google στην Ισπανία. Στην Γαλλία από ό,τι φαίνεται πέρασε ένας νόμος που ε, ασχολείται με το αποτύπωμα μικρές ε, εκδοχές φωτογραφιών σε αναζήτηση για τις φωτογραφίες και είπαν ότι θα υπάρχει πληρωμή, θα διανύμεται στους φωτογράφους μέσω μηχανών αναζήτησης ε, και προσπαθώ ακόμα να καταλάβω τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το νόμο και τι ανταπόκριση θα έχει. Σε γενικές γραμμές, νομίζω το 1999 όταν έγραφα για τα επιχειρήματα υπέρ της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και κάποιοι, φοβάμαι ε, και εγώ μεταξύ αυτών, αλλά δεν έχω ελέγξει τις πηγές, εξήγησαν ότι ένα βασικά από τα επιχειρήματα που εμφανίζονται εδώ στις Βρυξέλλες είναι ότι δεν θέλουμε αυτός ο οποίος παραδίδει το φάκελο που δίνει το ταχυδρομείο να είναι ο υπεύθυνο για τη δυσφήμιση εντός της του φακέλου. Επομένως, πρέπει να έχουμε αυτό το οποίο αποκαλείται στα Ηνωμένο, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, Safe Harbor ε, στις υπηρεσίες. Θα έπρεπε να είχαμε προσέξει πάρα πολύ την ερμηνεία αυτής της οδηγίας. Από ό,τι κατάλαβα, η Facebook και η Google είναι εκδότες. Κάποιος είπε, είπε ο Χάικο μας ε, τις προάλλες. Ίσως όπως έγινε με την AT&T στις Ηνωμένες Βολεσίες θα πρέπει να, ε, ε, να χωριστούν και να υπάρχει διάκριση μεταξύ της Facebook όταν τσανίκουν ε, οπτικές ίνες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού που δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τις οπτικούς ίνες και τι γίνεται με το Facebook ως εκδότη, ο, κυρίως ό,τι εκδίδει στην, στους των ανθρώπων και άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν χρήματα από τι εκδόσει αυτέ, θα ήταν μια καλή αρχή για να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο. Όσον αφορά του ισότιμους όρου, πραγματικά εγώ θα ήθελα να δω τι γίνεται με την αλυσίδα διανομή και κυρίω ισότιμους όρου μεταξύ εμού και των εκδοτών. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε Το να μου επιβάλλουν, για παράδειγμα, συμβόλαια και να θεωρείται παράνομο, παράνομο δεν μπορούν να το συσχετήσουν με τα όλα όσα συμβαίνουν. Ε, το να πληρώνουν βέβαια και οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις το φόρους, καλό θα ήταν. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητε. Πριν από κάποια χρόνια μελέτησα το μοντέλο στήριξη για τον τοπικό τύπο στη Σουηδία. Δεν είμαι όμω βέβαιος ε, κατά πόσον θα έχει αποτέλεσμα για ανθρώπου που δεν ζουν στη Σουηδία, σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα μέσα. Ε, ξεκινώ λοιπόν και πάω πίσω στην αρχική μου θέση, την οποία λέω και στους συναδέλφους. Να υπάρχουν ισότιμοι όρου για τους δημοσιογράφους ε, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες εφημερίδων και για τους ιδιοκτήτες εφημερίδων σε σχέση με τους ενδιαμέσους στο διαδίκτυο και ελπίζω ότι αυτά ε, θα γίνουν προς το συμφέρον της δημοκρατίας και ενός λογικού πολιτισμού και ότι θα μπορέσουμε έτσι να υποστηρίξουμε την έντυπη δημοσιογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. We uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας και γνωρίζουμε βεβαίως ε, ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η πρόκληση και πιστεύω ότι και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς με αυτό ασχολείται και αυτή η διάκριση μεταξύ εκδότη ή του διαμεσολαβητή, αυτού που παρέχει απλώς περιεχόμενο, είναι το βασικό ζήτημα. Και από νομική σκοπιά η λύση νομίζω ότι θα χρειαστεί βοήθεια. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και το περιεχόμενο και τους ορισμούς ε, και τις προσεγγίσεις, ε, διότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η πραγματικότητα. Φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Μετά θα ε, κάνουμε και τη συζήτηση βέβαια και θα ακούσουμε τι έχουν οι συνάδελφοι. Να δώσω τώρα το λόγο το, στο Σεμπάντια Ντέντεν, ιδιοκτήτη του Burta Media, ο οποίο θα ασχοληθεί κυρίω με μια εικόνα του τομέα της έντοπης δημοτιογραφίας για τους αναγνώστες και τη διαφήμιση και νομίζω ότι θα αναφερθεί και θα μας δώσετε και την άποψή σας για την ε, νομοθεσία που έχουμε ε, εξελίξει και για τα δικαιώματα του δημιουργού. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Um, I'm very pleased to have the opportunity. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να είμαι εδώ. Σήμερα σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που ήδη έθεσαν κάποια θέματα και χαίρομαι που εγώ τώρα παίρνω τώρα το λόγο. Εκπροσωπώ ήταν Hubert Burda Media, που είναι μια οικογενειακή μεγάλη επιχείρηση εντύπων με έδρα το Μόναχο, που απασχολεί 10.000 άτομα ανά τον κόσμο και έχει γύρω διαδικομαδιαδίες. Ίσως είναι οι, τους μεγαλύτερους εκδότες. Ε, εκδίδει 8 έντυπα στην ε, Γερμανία, το Focus, πολλά περιοδικά μόδα και πολλά ε, ε, έντυπα, στον, έντυπο, πάρα πολλά περιοδικά στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες και στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός το και το ψηφιακός ε, μέρος των πωλήσεων και ο έντυπος τύπος. Ξέρετε ότι έχουν γίνει και ε, διάφορες επενδύσεις ε, για άλλα τύπου περιοδικά σε άλλους τομείς στην D-Conferences Είχαμε και μία τέτοια διάσκεψη τον Δεκέμβριο και αυτό το πιο σημαντικό δικό μας ε, καινούργιο project είναι το Clicks, το οποίο εισαγάμε πρόσφατα στην αγορά και Βεβαίως ξέρουμε ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παίκτες. Αρχίζοντας θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον τίτλο κρίση στον έντυπο τύπο. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον εμείς δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως είναι, πρέπει να πω, ε, πολλές προκλήσεις σήμερα, όπως είπαν οι συναδελφοί, αλλά πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικός ο τομέας των ε, περιοδικών του έντυπου τύπου σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία. Βεβαίως αυτό δεν συμβαίνει για όλους. Υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν παρερμηνίες. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιους αριθμούς όσον αφορά και τα έσοδα τα οποία έχουμε και από την διαφήμιση, κυρίως στην Γερμανία. Αυτό στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο θα ήθελα να σας μιλήσω για διάφορα, ε, για την πρόταση για, ε, για την κοινοτική νομοθεσία και ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι όπως λέγεται το τον Microsoft το 2008, σε 10 χρόνια τα περιοδικά και ο έντυπος τύπος δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησε σε διάφορους λανθασμένους υπολογισμούς και η δική μας βιομηχανία στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ υγιής ακόμη. Κάθε χρόνο οι Γερμανοί αγοράζουν 2,5 δις περιοδικά συνολικού κόστους 260 εκατομμύρια κάθε μήνα και στην Μπούρτα εμείς πολλούμε περισσότερο από 300 εκατομμύρια περιοδικά ετησίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώ κατάσταση είναι. Αλλά βεβαίω, όπω καταλαβαίνετε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μια νέα κατάσταση στον τύπο και θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες εξελίξεις για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιε είναι οι ακριβείς αλλαγές και πώ ε, ε, χρειάζεται να ανταποκριθούμε και από πολιτική σκοπιά. Όπω είπε και ο συνάδελφος κατά παραδοσιακό τρόπο χρηματοδοτούνται τα περιοδικά από τις πωλήσει και από τα έσοδα που αποκομίζουμε από την διαφήμιση. σε αυτά διαφέρουν από έντυπο σε έντυπο. Ας δούμε τι γίνεται πρώτα απ' όλα στον τομέα των διαφημίσεων. Τα προηγούμενα 30 χρόνια το μερίδιο του τύπου στη Γερμανία μειώθηκε στον τομέα αυτό, από 29 έφτασε στο 30% για τις εφημερίδες και τα περιοδικά άλλα έντυπα. Αλλά κυρίως κατά την ίδια περίοδο πρέπει να πω ότι ε, τριπλασιάστηκε το μερίδιο της ε, τηλεόρασης, πράγμα που είναι αρκετά εκπληκτικό, εκπληκτικό διότι από ό,τι φαίνεται και σχετική οδηγία ε, δεν υφίσταται η τηλεόραση σχεδόν κανένα περιορισμό όσον αφορά την διαφήμιση. Και πιστεύουμε ότι δεν θα μας ε, ε βοηθήσει αυτό πάρα πολύ. Θα γνωρίζετε ίσως την μελέτη της Morgan Stanley, σύμφωνα με την οποία 85 cents κάθε δολαρίου που δαπανάτε για τη διαφήμιση ε, και επενδύεται στο ίντερνετ πηγαίνει σε δύο μεγάλες εταιρείες που τις γνωρίζουμε όλοι, την Google και την Facebook. Τώρα, οι αναγνώστες, πρέπει να πω οι δικοί μας τουλάχιστον, είναι πιστοί και χαίρονται διότι συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν και αγοράζουν πολλά περιοδικά. Ακόμη και όταν πρέπει να αυξήσουμε την ε, τιμή, την οποία αντιμετωπίζουν θετικά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ε, για τους εκδότες των εντύπων ε, αυτό, αυτή η αγορά είναι ένα μεγάλο πηγή εσόδων. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον για την δική μας την ε, βιομηχανία εντύπωση Γερμανία και δεν συμφωνούμε με τον τίτλο που λέει κρίση. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα, θα ήθελα να περάσω και στο πολιτικό σκέλος μάλλον της δικής μου της ε, παρέμβασης. Ε, ο ελεύθερος τύπος δεν ζητάει από τους πολιτικούς ούτε δώρα ούτε επιδόματα και βεβαίως πιστεύουμε ότι θα πρέπει σε κανονιστικό πλαίσιο να ενεργούμε όλοι ίσης όρης, να βρισκόμαστε δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με τους διεθνείς μας ανταγωνιστές. Πάρα πολλά έχουν ε, γίνει τους τελευταίους μήνες χάρη στην εργασία που έχει επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να πω ότι η Ευρώπη έχει κάνει ε, πολλά βήματα προς την εξασφάλιση ίσων ε, δυνατοτήτων για όλους σε τομείς πολύ σημαντικούς όπως η προστασία των δεδομένων, η φορολογία, η αντιμονοπωλιακή πολιτική και Ξέρετε τι ε, ακριβώς λέγεται για τα ψηφιακά μονοπολία. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ως εκπρόσωποι εκδοτικών οίκων ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο ώστε όλοι να χαίρουν των ε, ιδίων ε, ε, όρων στην αγορά. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί στόχοι θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη να μπορούν σε μια κοινωνία που λειτουργεί σωστά να επιτρέπουμε σε όλους να συμμετέχουν. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η στριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων εργάζονται για εκδοτικούς οίκους. Στη Γερμανία τουλάχιστον περίπου τα δύο τρίτα αυτών. Και από παρά τις διάφορες προβλέψεις από τη δεκαετία του 90, οι bloggers και οι αυτοί που, κάνουν, ε, που είναι μόνοι και ενεργούν και κάνουν ε, την διαφήμιση δεν έχουν ε, υπεσκελίσει τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Βεβαίως όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο κόστος κάποιος, ε, κάποιο κόστος για τους ε, επαγγελματίες δημοσιογράφους και διότι που ε, θέλουν πραγματικά να παρέχουν πληροφορίες αξιόπιστες. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ποιότητα στην ενημέρωση και δαπάνες οικονομικές για τους εκδότες. Σας έδωσε διάφορα στοιχεία ο συνάδελφος σε σχέση με αυτό. Επίσης, το θέμα της αναχρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι είναι αυτό ένα δύσκολο ε, θέμα ε, να αντιμετωπιστεί. Είναι πάρα πολλά ε, περιεχόμενα ελεύθερα και είναι δύσκολο κανείς να μπορέσει να βρει το σωστό. Βεβαίω επίσης υπάρχει από την άλλη ο ψηφιακός κόσμος, υπάρχει υπεραυθονία ε, χώρου για διαφήμιση στο ίντερνετ. Κάποιο άλλο το οποίο είναι χαρακτηριστικό από την εποχή που άρχισε να χρησιμοποιήσει τον, ε, η ψηφιοποίηση και τον ίντερνετ είναι οι νέοι μεσάζοντες οι οποίοι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή διάφορες μηχανές αναζήτησης, φορείς που συγκεντρώνουν τα διαδικτυακά εργαλεία. Πολλοί αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, πράγμα το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στην ε, στους χρήστες και όπως σας είπα πώς επενδύονται 85 εκατοστά του κάθε νέου δολαρίου που επενδύεται στην ε, διαφήμιση online και επικεντρώνεται σε δύο εταιρείες μόνο την Google και την Facebook και βεβαίως σε όλη τη διαδικασία λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι εποφελούνται από όλα αυτά τα κέρδη και από τους ε, ε μεσάζοντες οι οποίοι όπως σας είπα επικεντρώνονται. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία να κερδίζουν οι πάντες αλλά Βασικά μέχρι τώρα τα πράγματα στον τομέα αυτό είναι ασυμμετρικά και άδικα. Άρα η πρόθεσή μας είναι να μπορέσουμε στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού να κάνουμε ε, διάφορες ε, ε, συμφωνίες οι οποίες ε, θα είναι θετικές και υποφελείς για όλους. Χρειάζεται όμως να έχουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο κυρίως για να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα όλων των προϊόντων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόταση της Επιτροπής πηγαίνει προς την ε, σωστή κατεύθυνση και στην Γερμανία πρέπει να σας πω ότι έχουμε από καιρό αντιμετωπίσει το όλο θέμα. Τα έχουμε μάθει πώς λειτουργούν τα πράγματα, κυρίως και σε σχέση με την δική μας την νομοθεσία και για να μην υπάρχουν αρνητικά σενάρια, πιστεύουμε ότι θα πρέπει πραγματικά ο Ευρωπαίος νομοθέτης να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην αναπτύσσονται περαιτέρω μονοπωλιακές πλαθόνες και να υπάρχει σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι ίσως κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλει κάποιος να ζητήσει περισσότερο λεπτομέρειες. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν παρανομηθεί. Πρώτα απ' όλα, ότι ε, το, ε, οι διάφοροι εκδότες θέλουν να συνδέσουν την πρόσβαση στους διάφορους συνδέσμους, σε διάφορα link τους με χρήμα. Επίσης ότι θέλουμε να μπλοκάρουμε κάποια περιεχόμενα και αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα και αυτά. Νομίζω ότι ετέθησαν πολλά θέματα επιτάπητος και νομίζω ότι από όλε τι ε, παρουσιάσεις ε, προκύπτει σίγουρα το εξή. Εσείς είπατε ότι δεν υπάρχει κρίση διότι τα στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι υπάρχει μια τροποποίηση και του χρήστη. Υπάρχει αλλαγή λοιπόν στη συμπεριφορά ε, λόγω της ψηφιακής εξέλιξης, αλλά μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη δίψα για περιεχόμενο και για πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά και οι τρεις νομίζω ότι προβάλλατε σαφέστατα ότι χωρίς ένα κατάλληλο πλαίσιο, είτε σε νομιθετικό επίπεδο, είτε σε πλαίσιο ισότιμων όρων, αυτή η πιθανή ανάπτυξη και από πλευράς ε, του χρήστη και από πλευράς ε, της προσφοράς ε, θα πρέπει να γίνει με θεμητούς όρους ε, και επομένως και η έντυπη δημοσιογραφία θα πρέπει να έχει το χώρο της μέσα σε όλο αυτό το ε, πανόραμα των μέσων ενημέρωσης. Και κάτι άλλο το οποίο ε, αναφέρατε είναι η ποιότητα του περιεχομένου πέραν της πολυφωνίας της πληροφορίας που πρέπει να παραμείνει διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει και ε, επένδυση από πλευράς εκδοτικών οίκων ε, σε επαγγελματίες δημοσιογράφους που είναι πολύ σημαντικό που μας είπατε κι εσείς ότι αυτή είναι στο επίκεντρο. Η πρόσβαση στους πόρους λοιπόν και η επαλήθευση των πόρων γίνεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε δημοκρατικό επίπεδο. Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα για μας. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν το οποίο μας παρουσιάσατε κι εσείς της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε την αποκλειστική αρμοδιότητα εμείς ως αρμόδια επιτροπή για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε και τους δύο εισηγητές και τους και όδης εδώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Επιτροπή μας ε, και τα εξετάσαμε λοιπόν όλα αυτά και για την ψηφιακή στρατηγική. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Φερχάιεν και μετά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαλτέζε γιατί αυτός ε, έκανε την πρόταση, στην Τζούλι Γουόρτ και στην Χελγα Τρούπελ. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, τρει ομιλητέ. Πιστεύω πως μας δώσατε μία πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στον κλάδο αυτήν την εποχή, τι γίνεται με τους ε, δημοσιογράφου και μας δώσατε επίσης και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα ε, μιλώντας και για την νομοθεσία που διαθέτει ε, νομίζω όμως πως έχουν παραμείνει ανοιχτά κάποια ερωτήματα. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των ε, δημοσιογραφικών οργανώσεων το ε, τι σημαίνει ακριβώς η, η θεμητό ανταγωνισμό για του ε, δημοσιογράφου. Ξέρω πω τα τελευταία χρόνια απολύθηκαν πολλοί δημοσιογράφοι, αντικαταστάθηκαν από ελεύθερου επαγγελματίε, κοστίζουν λιγότερο, δεν υπάρχουν λοιπόν ε, συμβόλαια αφού μειώθηκαν αυτές οι θέσεις. Μπορούμε να πούμε επομένως πως ε, υπάρχει μια κρίση ε, στον δημοσιογραφικό κλάδο. Αυτό συνδέεται και με μια απώλεια όχι μόνο θέσεων απασχόλησης αλλά και ποιότητας ακριβώς επειδή στους ε, εκδοτικούς οίκους έχει μειωθεί το προσωπικό, απασχολούνται οι ε, δημοσιογράφοι ή μάλιστα όσοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους έχουν αναλάβει καθήκοντα πολύ περισσότερα από όσα είχαν. Πώς μπορούμε να το ε, αναλύσουμε αυτό ιδιαίτερα και τι συμβαίνει στις ε, τοπικές εφημερίδες, τα τοπικά περιοδικά αυτό επίσης συνδέεται και με κάποιο δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει. Πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, ε, την κάλυψη των ε, μικρών των ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό μπορείτε να το απαντήσετε όποιος από εσάς επιθυμεί, όποιος από τους δύο. Μετά μας είπατε για πηγή εσόδων για τα έντυπα μέσα, τις διαφημίσεις δηλαδή. Πώς ε, υπάρχουν διάφορες ε, μορφές ε, διαφημίσεων, διάφορες μορφές εσόδων, πως έχουν χαθεί τα παραδοσιακά έσοδα από τις διαφημίσεις. Αυτή τη στιγμή πολλοί εκδοτικοί οίκοι έχουν και ε, παρουσία στο διαδίκτυο, έχουν επιγραμμική πλατφόρμα, προτιμούν λοιπόν να διοχετεύσουν τις διαφημίσεις και τη χρηματοδότησή τους εκεί. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές, τελείως ανεξάρτητες διαφημίσεις οι οποίες τοποθετούνται μόνο στο διαδίκτυο δεν, ε, και τα έσοδα δεν διοχετεύονται και στα έντυπα μέσα ενός εκδοτικού οικού. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντισταθμίσουμε αυτήν την απώλεια εσόδων έτσι ώστε να μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικά τα έντυπα μέσα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, κρίσιμο ερώτημα και θα ήθελα να μάθω τις αντιδράσεις του κλάδου, τις αντιδράσεις των εκδοτικών οίκων σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, στο θέμα του ΦΠΑ, νομίζω πως συμφωνούμε οι περισσότεροι εδώ ότι τα επιγραμμικά προϊόντα, τα αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν διαφορετικό φορολογικό συντελεστή από τα έντυπα. Νομίζω πως είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν άλλωστε. Ε, τώρα, όσον, σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, νομίζω πως ε, χρειάζεται αποτελεσματική δράση. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση από το να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι πάροχοι των υπηρεσιών μαζί, μουσική, βιβλία, οι ηλεκτρονικές εκδόσει πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ε, ίδιε υποχρεώσεις. Είτε αυτό είναι περιοδικό τύπος, είτε αυτό είναι διαδικτυακό. Εσείς έχετε όμως ε, να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Νομίζω πως στη Γερμανία έχει γίνει ήδη μία προσπάθεια από τους ε, εκδοτικούς οίκους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, να αντιμετωπίσουν το μονοπόλιο που έχει δημιουργηθεί από αυτές τις ε, δύο-τρεις εταιρείες. Πώς μπορούμε όμως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες και να διευκολύνουμε έτσι την ε, επιβίωση αυτών των εκδοτικών οίκων, να διευκολύνουμε την επιβίωση της ελευθεροτυπίας. Χρειάζεται αποτελεσματική νομοθεσία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη, τους ε, μεσάζοντες ή τις ε, συγκεντρωτικές πλατφόρμες ε, ειδήσεων. Και χρειάζεται βέβαια αυτή η λύση να είναι αναλογική και να ε, πληρώνει περισσότερο αυτός που ε, συγκεντρώνει περισσότερες διαφημίσεις, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο συνάδελφο Μαλτέζε. Ναι, εγώ είμαι δημοσιογράφο εδώ και 35 χρόνια, από τότε που ήμουν νεαρό. Ε, και σε μεγάλες εφημερίδες, οι οποίες ήταν πάντα ε, ενεργές και μου επέτρεπαν να ασκώ σωστά τη δημοσιογραφία μου. Ε, κέρδιζα καλά λεφτά και κέρδιζε και ο εκδότης μου. Και ο εκδότης μου χαιρόταν που κέρδιζε και έτσι μ' άφηνε να γράφω και πράγματα πολύ διαφορετικά από τη δική του την άποψη, αν θέλετε. Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να είναι δημοσιογράφος με αυτή την έννοια. Αυτό είναι γεγονός. Το διαδίκτυο άλλαξε τα πάντα. Και πλέον δεν γνωρίζουμε πολύ καλά πώς τα άλλαξε. Ξέρουμε ότι για δύο αιώνες ο ρόλος της γραπτής ενημέρωσης στη δημοκρατία ήταν πάρα πολύ σημαντικός κυρίως όταν απευθύνεται με λογικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση. Σήμερα τα νέα μέσα απευθύνονται με παράλογο κυρίως τρόπο ε, στην ε, ε, δημοκρατία και αυτό είναι και μια διαπίστωση. Αλλά βρισκόμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως νομοθέτες. Διότι Αφενός υπάρχει εντύπωση ότι οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν αυτό το μεταβατικό στάδιο για να μπορέσουν να αφαιρέσουν δικαιώματα από τους δημοσιογράφους, κυρίως από τους νέους δημοσιογράφους και δεν υπάρχει απλώς μια επανάσταση εν εξελίξη, αλλά υπάρχει και η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί αυτή η επανάσταση για να μειωθεί ο χώρος της αυτονομίας όποιου ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αυτό είναι σαφές και στην οικονομική κατάσταση στην οποία υποχρεώνονται να εργάζονται αυτοί οι νέοι και στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες κλπ. Επίσης υπάρχει ένα νομοθετικό κενό πολύ σημαντικό ε, λίγο γιατί είναι δύσκολο να νομοθετήσει κάποιος ε, για ένα σύμπαν το οποίο αλλάζει τόσο γρήγορα. Και λίγο και γιατί δεν ε, επιθυμούμε κιόλας να το κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν το 85% των πόρων της διαφήμισης να καταλήγουν στα χέρια της Google και της Facebook. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουν και φόρους η Google και η Facebook όταν πρέπει να πληρώνουν. Και επίσης δεν είναι δυνατόν να είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο το οποίο κυκλοφορεί. Εάν εγώ είμαι εκδότης σε μια εφημερίδα, ενό περιοδικού, είμαι υπεύθυνο και για αυτά τα οποία γράφονται στις επιστολές που δημοσιεύω εγώ που έχουν γράψει αναγνώστε. Εάν εγώ λοιπόν είμαι υπεύθυνο για το YouTube ή για οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία μοιράζεται περιεχόμενο, δεν είμαι υπεύθυνο για τίποτα. Ένα άρθρο δικό μου, το οποίο έχω γράψει εγώ στη Ρεπούμπλικα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, ε, μπορεί ε, να δια... έχει σχέση για μένα, αν εγώ καταδικαστώ, μπορεί να καταδικαστώ εξαιτία του άρθρου. Αν αυτό το άρθρο το χρησιμοποιήσει κάποιος στο facebook, δεν συμβαίνει τίποτα ε, και βρίσκομαι στο απειρόβλητο. Αυτό στην πραγματικότητα ε, είναι αντικειμενική βοήθεια για να αναδυθεί η χειρότερη δυνατή οδός προς τις νέες τεχνολογίες. Διότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ε, δραματικά η δημοκρατία. Και ε, όσον αφορά τους οικονομικούς υπολογισμούς, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κανένας ε, στο χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας δεν πιστεύει ότι τα αντίγραφα της Frankfurter Allgemeiner είναι τα ίδια με τις Bild ή ότι η Ρεπούμπλικα είναι αντίστοιχη μιας εφημερίδες ε, άλλου επίπεδου. Και το αυτό φυσικά ισχύει και για άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γιατί στο διαδίκτυο δεν γίνεται διάκριση στους υπολογισμούς ε, και στη διαφήμιση. Αν ένας αναγνώστης διαβάσει ένα ραπορτάζ 10 σελίδων για το Ιράν ή για την ευρωπαϊκή πολιτική, δεν είναι το ίδιο με κάποιον ο οποίος ε, ε, θα δει τις Playmate του μήνα σε 50 φωτογραφίες. Ε, και αυτά μετρούνται με τον ίδιο τρόπο. Και από πλευράς διαφημιστικής ε, είναι τελείως διαφορετική η προσοχή και οι αγορές στις οποίες επικεντρωνόμαστε είναι τελείως διαφορετικές. Αυτό στην έντυπη δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η ποιότητα δεν ανταποκρίνεται στην ποσότητα και η ποσότητα δεν είναι πιο σημαντική από την προσοχή που αφιερώνει το κοινό στο περιεχόμενο και στο προϊόν. Ευχαριστώ Κούρτσιο, όπως βλέπετε είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και θεωρώ ότι πρέπει να τα σκεφτούμε από κοινού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και από πλευρά ποιότητα και από πλευρά ελευθερία και δημοκρατία, όχι μόνο για το έργο των δημοσιογράφων. Τώρα θα δώσω το λόγο στη Ζούλη Γουόλτ και μετά στην Μιχαήλ Κατρούπολη. Um, thank you for... Ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συζητούμε αυτό το θέμα εδώ σήμερα. Άκουσα με χαρά την, ε, αυτά που για την... Πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ηθικής στην εργασία, στις επιχειρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο και σε επίπεδο παιδείας. Θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύω ότι είναι πραγματικής ε, σημασίας για μας να είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι και δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν όλοι οι νέοι να αναρωτιούνται αν αυτά τα οποία διαβάζουν είναι σωστά και ε, ακόμη και να θέτουν σε αμφισβήτηση διάφορες ακραίες παρουσιάσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας ε, με την ε, θλιβερό γεγονός της δολοφονίας της Τζο Κόξ Βεβαίως, δεν θα πω ότι στις εφημερίδες δεν προωθήθηκαν κατά κόρον ακραίες θέσεις για χρόνια και κυρίως διάφορα σχόλια αρνητικά για το θέμα του δημοψηφίσματος, αλλά για το πώς συνδέεται αυτό το γεγονός με αυτή τη δομή. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ ε, μελετήσει θέματα που αφορούν τον πολίτη, την κοινωνία στην οποία ζει, την δημοκρατία, τέτοιου είδους θέματα, να τα πραγματεύεται, να τα εξετάζετε σωστά ο τύπος. Πρέπει να σας πω ότι στην Ολλανδία, από ό,τι ξέρω, γίνεται μία πάρα πολύ σημαντική δουλειά με τα παιδιά, ε, τα οποία πρέπει γίνεται προσπάθεια να συναντήσουν τους ε, εκλεγμένους εκπροσώπους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, να, να κατανοήσουν και εμείς τι ακριβώς κάνουμε και εμείς τι κάνουν εκείνοι. Πριν να ε, ασχοληθώ με την πολιτική, πρέπει να σας πω ότι ασχολήθηκα με την ε, τέχνη και τα μέσα τα σχετικά. Και υπήρχε σχέδιο διασύνδεσης μίας ε, ε, περίπτωση που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με το πώς θα με το, να παρακολουθήσουν μια τέτοιο είδους δίκη νέοι και να μπορέσουν να την σχολιάσουν και να τη συζητήσουν μετά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μας είπαν σήμερα οι δημοσιογράφοι μας ότι υπάρχει ενθουσιασμός μεταξύ των νέων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, όπου υπάρχει κενό για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων να το να ασχοληθούν και να πληρώσουν αυτό το κενό. Νομίζω ότι υπάρχει σε εσά μεγάλο ε, βάρος αλλά θετικό για να μπορέσετε αυτά τα οποία τα κενά που υπάρχουν να τα πληρώσετε για να ανταποκριθούμε σε προβλήματα τα οποία έχουν ε, τα ε, νέα παιδιά. Um, an issue that really concerns me, which is the distribution of free newspapers Επίσης, τα θέματα της ε, ε σωστής πληροφόρησης και σε ποιος πρέπει να ηγείται των διαφόρων. πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, με την ακραίες, ακραία ε, δεξιές θέσεις και ακραίες θέσεις που παρουσιάζονται ε, Υπάρχουν προσπάθειες από τον τύπο να προσεγγίσουν το καθένα, ακόμη και με έντυπα τα οποία ε, στέλνουν στο σπίτι, δέδοντας ε, και ε, ελεύθερα μοιράζοντας έντυπα και εφημερίδες και κυρίως εκμεταλλεύονται διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις. Τελικά, υπάρχει το εξή θέμα. Τι γίνεται τώρα με τους δημοσιογράφους στην Τουρκία. Οι Κούρδοι βεβαίως όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο ή με τους υπόλοιπους ε, Κούρδους εκτός Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχουν φημωθεί αυτή τη στιγμή η δημοσιογράφος. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται. Η γνώση και η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτοί οι δημοσιογράφοι διότι δεν μπορούν να πούνε την αλήθεια και είναι επικίνδυνοι για την επίσημη κυβέρνηση του κράτους αυτού. Ευχαριστώ. Η ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις που έκαναν οι προσκεκλημένοι μας. Όταν δημοσίευσε η Επιτροπή της Προτάσης για την αναθεώρηση των πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να σας πω ότι έγινα επικριτική για τα... Ε, δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν των υστέρων και οι εκδοτικοί. Εσείς το αναφέρατε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνετε τώρα με απόλυτη σαφήνεια είναι να δείτε πώς μπορούν πώς μπορείτε να ε, καθορίσετε τον ε, ρόλο των ε, ενδιαμέσων, των μεσαζώνων και να κάνετε πάρα πολύ καλή, καλό διαχωρισμό και ορισμό μεταξύ εκδοτών, εντύπων και αυτών. Θα πρέπει λοιπόν εσείς να δείτε κατά πόσον διαφοροποιείται ο ρόλος τους. Επίσης, βλέπουμε στον τομέα αυτό το γενικό πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει. Όλοι θέλουν να έχουν ελεύθερο ίντερνετ, απ' την άλλη όμως πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλό ε, νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε το μονοπόλιο του ίντερνετ. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο σκέλη της πολιτικής. Από πολιτικής πλευράς είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Όπως είπα και στην πρώτη μου ερώτηση, πώς νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τον διαχωρισμό, πώς μπορείτε ε, ε, να μας πείτε ποια είναι η αναλογία μεταξύ των δύο προτάσεων. Επίσης, υπήρχε μία, το κριτική που έγινε πριν από 10 χρόνια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπήρχαν διάφορε παρεμφερεί εκδόσει εφημερίδων στον, ψηφια, στον ε, αναλογικό μας ε, κόσμο πριν εμφανιστεί το ίντερνετ. Για μένα αυτό είναι μέρος του προβλήματος, διότι βεβαίω, και έχει, και έχει αυτό σχέση με την συμπεριφορά των διαφόρων ε, μεσαζόντων, των διαμέσων. Ένα από τα, άλλα προβλήματα ήταν, από προβλήματα είναι ότι όλα τα περιεχόμενα που έχουμε σήμερα σχεδόν είναι, ε, παρέχονται δωρεάν. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Και για τον κύριο Χόλντενερ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την πρόταση της Επιτροπής για αυτά τα επικουρικά ε, και δευτερεύοντα πνευματικά δικαιώματα. Πώς ε, βρίσκεται την πρόταση αυτή. Θέλετε να ε, προσθέσετε κάτι, την φοβούνται οι δημοσιογράφοι. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αναλογία και μερίδιο μεταξύ όλων των εκδοτών και των ε, μέσα ζώνων. Αλλά βεβαίως πρέπει να πω ότι ο γερμανικός νόμος, η γερμανική νομοθεσία δεν ήταν ε, ιδιαίτερα υποφελής κυρίως για τους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρώτα θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτον, ε, το θέμα αυτό με βρίσκει σύμφωνη, συμφωνώ και με αυτά που είπαν αρκετοί συνάδελφοι και θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κατά πόσον η προσέγγισή σας ε, για το θέμα αυτό, ε, με την οποία συμφωνώ, να βρούμε νέους τρόπους να είναι υπεύθυνε οι διάφορες πλατφόρμες και γι' αυτό είχαμε και μια συγκεκριμένη πρόταση ως ε, Ένωση των Εκδοτών, ε, το σεβασμό, για παράδειγμα, ε, της ευθύνης των εκδοτών. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ε, οι εκδότες είναι υπεύθυνοι και όταν οργανώνουν και όταν επιλέγουν κάποια θέματα και κυρίως πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τα, το αντίστοιχο θέμα στο διαδίκτυο. Και οι συγγήτριες λοιπόν είναι κάτι που τους απασχολεί. Είναι ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί αρκετά και δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίως όμως όταν ανδιαφερθήκαμε σε δύο πτυχές, εκεί είχαμε κάτι καλύτερο. Τη δυνατότητα να υπάρχουν μεγαλύτερες ευθύνες ε, ε, για τις πλατφόρμες, για παράδειγμα, που μοιράζονται ε, βίντεο σε θέματα προστασίας των ανηλίκων και hate speech, ε, αλλά ε, για τα άλλα θέματα δεν είχαμε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και ο κύριος Χόλτερνες μας είπε, ο κύριος Ντόντεν, συγγνώμη, μας είπε ότι δεν αντιμετωπίζει κρίση η έντυπη δημοσιογραφία αλλά υπάρχει κρίση των δημοσιογράφων, υπάρχει θέμα ανταγωνισμών που δεν θα έπρεπε όμως να γίνει για τις εφημερίδες ε, ανταγωνισμός προς τα κάτω, δηλαδή να μην επενδύουν ε, ε, σε επαγγελματίες, διότι θα υπάρχει ανισότητα και για την έντυπη δημοσιογραφία. αλλά και το περιεχόμενο στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή ε, έχουν θέμα ποιότητας ε, και αν είναι ψηλό ο ανταγωνισμός ε, μπορεί να προσφερθεί και σε διαδικτυακό επίπεδο. Μήπως υπάρχει μια αντίφαση λοιπόν εδώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο Τζορέλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής θυματιάρχης του τμήματος ε, για τα πνευματικά δικαιώματα της Γενικής Διεύθυνσης Κονέκ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. κάποια ε, στοιχεία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η συζήτηση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, αυτό το οποίο κάνουμε δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Connect και κυρίως τις προτάσεις που μόλις ε, καταθέσαμε για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, βρισκόμαστε βεβαίως στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας. θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως για τα πνευματικά δικαιώματα, να γίνουν πιο διεξοδικές συζητήσεις κάποια στοιχεία, όπως σας είπα, θα σας δώσω σήμερα. Αναφέρθηκε ήδη και από τους ομιλητές ότι και η διάσταση των εκδοτών και των ε, συντακτών ε, ως δημιουργοί και ως άνθρωποι που επενδύουν, επενδύουν στη δημιουργία της ποιοτικής δημοσιογραφίας είναι στο επίκεντρο της ε, ε, πολιτικής μας για τα μέσα και της πρόσφατης ε, πρότασής μας ε, για τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένας τομέας στον οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και είναι ίσως και το πιο ε, καινούριο κομμάτι των προτάσεων για τα πνευματικά δικαιώματα. Το πιο καινούριο με την έννοια ότι ε, κάποιοι άλλοι τομεί ε, της δέσμης μέτρων είναι απλώς μια επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου. Εδώ προσπαθούμε να πάμε λίγο περισσότερο και να ε, ανοίξουμε νέες δυνατότητες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι στο παρόν οικοσύστημα, στην ε, παρούσα οικονομία του διαδικτύου, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πνευματικά δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούν να υποστηρίξουν ε, τις επενδύσεις στη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου. Ε, βέβαια, ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το ε, δικαίωμα γειτονία αυτό το neighboring right και επίσης δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τις εφημερίδες ή τους εκδότες, θέλουμε να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις στη δημιουργία περιεχομένου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιτρέψει να εξηγήσουμε και από πού ξεκινήσαμε. στην πρόταση έχουμε κάτι το οποίο υπάρχει ήδη σε άλλους τομείς ε, της δημιουργικής βιομηχανίας. Υπάρχει το λεγόμενο σχετικό δικαίωμα, related right. Πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο ανατίθεται στους εκδότες ως αυτούς οι οποίοι επενδύουν στο περιεχόμενο και αφορά και τα δικαιώματα των ε, ε, συντακτών, των δημοσιογράφων που όπως είπαμε ε, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται καθόλου και δεν επηρεάζονται καθόλου από την πρόταση και την εισαγωγή αυτού του neighboring rights. Και αποφασίσαμε να υποβάλουμε αυτή την πρόταση, εν μέρη γιατί υπάρχει εμπειρία της Ισπανίας και της Γερμανίας, οι οποίες κατά την άποψή μας ε, έχουν κάτι διαφορετικό. Η Ισπανική και η Γερμανική νομοθεσία είναι κάτι διαφορετικό από τεχνική σκοπιά από αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αποφασίσαμε να υποβάλουμε αυτή την πρόταση για να λάβουμε υπόψη το συγκεκριμένο ρόλο του τύπου στο διαδίκτυο. Και νομίζω ότι εν τέλει αυτό το οποίο συζητούμε εδώ είναι ότι με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη του διαδικτύου διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία χρήση υπό την έννοια του αγαθού. Ε, έτσι είναι το έντυπο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα με την οποία ε, χρησιμοποιείται το περιεχόμενο των εφημερίδων και αυτό δεν είναι μόνο θέμα των αλλαγών, αλλά γενικότερα. Υπάρχουν αρκετοί παρόχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ε, περιεχόμενο εφημερίδων σε μια γκρίζα ζώνη συχνά χρησιμοποιούν αποσπάσματα, κομματάκια, κάνουν ξανά συναρμολόγηση ενός κειμένου και κάτι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένο και γίνεται με την παροχή ε, περιεχομένου εφημερίδων στο διαδίκτυο. Ε, αναφέρθηκε ήδη, αλλά το διευκρινίσαμε και εμείς, ελπίζουμε στην πρόταση ότι δεν ε, αφορά ε, το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επηρεάζει το πεδίο εφαρμογή αυτού του οποίου καλύπτεται ή δεν καλύπτεται από τα πνευματικά δικαιώματα. Από πλευρά, για παράδειγμα, τη συζήτηση για, τα παρα, ε, για τις παραπομπές. Ε, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που καλύπτει τα θέματα αυτά. Το κατά πόσον, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιείς κάποιος ένα απόσπασμα κάποιου ε, ε, και πώς καλύπτεται και τι θεωρείται πνευματικό δικαιώμα εκεί. Αυτό έχει καλυφθεί ήδη από την νομοθεσία, δεν το επιτυράζουμε εμείς την πρόταση. Τώρα το κατά πόσον η πρόταση είναι καινούργια εντελώς, ε, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποιες επικρίσεις οι οποίες ε, αφορούν ε, τη χρήση του hyperlinking και κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν στη συζήτηση. Ε, είναι κάτι βέβαια το οποίο θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω για το Neighboring Rights, κατά την άποψή μας πρόκειται για μια τελείως διαφορετική συζήτηση σε σχέση με τη συζήτηση από την απαλλαγή της ευθύνη των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί τρόπον την να να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση για άλλα μέτρα τα οποία έχουν ε, ε, υποβληθεί για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά όχι τόσο για τη χρήση του περιεχομένου των εφημερίδων στο διαδίκτυο. Ε, δεν έχω ακούσει ποτέ, για παράδειγμα, να θεωρεί Google News ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο μιας εφημερίας, εφημερίδας ε, στο διαδίκτυο λόγω εξαιρέσεων στον τομέα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λίγο διαφορετική συζήτηση. Η συζήτηση είναι περισσότερο οι προϋποθέσεις με τις οποίες ε, περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο των εφημερίδων θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο επί τη βάση ε, πρώτερης άδειας ε, των εκδοτών. Όπως είπα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ε, περισσότερο στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος πολιτικής, ο οποίος πηγαίνει πέραν της συγκεκριμένη κατάστασης των εκδοτών των εφημερίδων και αφορά την ε, προστασία των επενδύσεων. Νομίζω για τα πνευματικά δικαιώματα θα μπορούσα να σταματήσω εδώ μία παρατήρηση ακόμα έγινε για την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες ε, και την ιδέα ότι οι νέοι κανόνες που προτάθηκαν για τη χρήση διαφημίσεων από ως μεταδίδουν περιεχόμενο θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά ε, τον κλάδο των εφημερίδων. Δεν πιστεύουμε ότι ισχύει αυτό, διότι υπάρχει ο κανόνας του 20% ορίου στις διαφημίσεις, ο οποίος άλλαξε τώρα με τρόπο ε, που θα επιτρέπει να υπάρχει διαφορετική καλύτερη κατανομή των διαφημίσεων στη διάρκεια της ημέρας, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των διαφημίσεων που μπορούν να κάνουν όσοι μεταδίδουν περιεχόμενο ε, τηλεοπτικό για παράδειγμα. Επομένως δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τις εφημερίδες γιατί δεν τίφτε θέμα ανταγωνισμού στη διαφημιστική πίτα. Ε, αυτό βέβαια ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να το ε, εξηγήσουμε και στο παρελθόν. Αυτά νομίζω. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα και σίγουρα θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε. Κυρίως για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Κύριε Χόλτενες, έχετε το λόγο. Ναι, θέλω μια ώρα για να απαντήσω. Κάπου τόσο υπολογίζω. Εντάξει, αστείευομαι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Τώρα, αντίστροφη σειρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν. Να πω καταρχάς ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη γερμανική νομοθεσία, κυρία Τρούπελ, είναι πως ε, δεν έγιναν ε, σαφείς οι διατάξεις για πληρωμές των δημοσιογράφων. Ε, τώρα, είπατε πως πρέπει να ε, στηρίξουμε τις επενδύσεις. Φυσικά, γίνονται επενδύσεις σε χρόνο, χρόνια ε, που ξοδεύει ένας δημοσιογράφος με ελάχιστες απολαβές για να αποκτήσει φήμη. Όταν είσαι όμως ελεύθερος επαγγελματίας μπορείς να γράψεις ένα άρθρο και να πας σε κάποιον να τον ρωτήσεις θες να το δημοσιεύσεις, σου αρέσει. Αυτό είναι μια επένδυση θεωρητικά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα επηρεάσει, ε, λέτε, τα δικαιώματα του δημιουργού. Η πρόταση το λέει αυτό, όμως αυτό προβλέπεται και από το ε, Διεθνές Δίκαιο για τα δικαιώματα των μουσικών παραγωγών σε, μια, σε ένα εχογραφημένο κομμάτι. Φυσικά βέβαια όταν πρόκειται για μουσική πρέπει να πας να βρεις αυτόν που έχει ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό προτού μιλήσεις στον δημιουργό, στο συνθέτη, στη χορό κτλ. Ε, αυτό ονομάζεται gatekeeper effect. Υπάρχει δηλαδή μια λασιδωτή αντίδραση όπου αυτά τα συγγενικά δικαιώματα θεωρητικά προστατεύοντας την πράξη όμως ε, τα πράγματα είναι αλλιώς. Στην ουσία δηλαδή τι γίνεται. Εσείς μας λέτε πως πρέπει να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο για να ε, πολεμήσουμε τα μονοπόλια. Αυτό όμως ε, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να είναι έξυπνος τρόπος, πρέπει να είναι σαφέστατος. Χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς κανόνες για το πού θα πηγαίνουν τα έσοδα, για το ποιος θα είναι ο δικαιούχος. Κυρία Ward. διανομή μας είπατε στο Λίβερπουλ. Τι σαν, ε, περίεργο μου φαίνεται, χαζό μου φαίνεται, σωματοφύλακες ε, χρειάζεται για να γίνει αυτό μας ε, είπατε κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω πως αφορά συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, πληροφοριοδότες, ε, θα υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίζουν ένα δημοσιογράφο, να του δίνουν εμπιστευτικέ και απόλυτες πληροφορίες, χωρίς να ε, αναγκαία να θέτουν σε κίνδυνο την υπόλοιψή του, την καριέρα του, τη ζωή του σε πολλέ περιπτώσεις. Ε, με ανησυχεί όμω πάρα πολύ ο νόμος που ψηφίστηκε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο σχετικά με ε, τις με τις ε, υποκλοπές πληροφοριών. Και η Αρμόδια Επιτροπή Διοντολογία στο Cambridge ε, έχει αποφανθεί ότι ε, όσον αφορά τους πληροφοριοδότες είναι σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να επιστρέψουμε στην παλαιόλιθική εποχή. Τι θα κάνουμε. με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι μεγάλα τα προβλήματα. Κάποιο δηλαδή πληροφοριοδότη θα θεωρηθεί πω είναι εγκληματία γιατί έχει υποκλέψει πληροφορίε. Τώρα, εκπαίδευση. Ναι, στα σχολεία χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που έχει αποδειχθεί αρκετά δημοφιλέ σε αρκετές χώρες. Κύριε Μαλτέζε, δυστυχώς έφυγε ο κύριος Μαλτέζε. Ευχαριστώ όμω πολύ, έστω και από μακριά, συμφωνώ με όσα είπατε. Κυρία Φερχάιεν. Η ερώτησή σας αφορά την, ε, την ε, μείωση της ποιότητας. Βέβαια η δική μου θέση είναι πολύ διαφορετική από του συνάδελφου δίπλα που εκπροσωπεί τον εκδοτικό οίκο Αλλά θα μπορούσα εγώ να πω πως ε, έχουν πληγεί πάρα πολύ τα μικρά μέσα ενημέρωση σε αντίθεση με τα μεγάλα. όλο το νότιο Λονδίνο, εκεί όπου εδρεύουν δηλαδή περισσότεροι δημοσιογράφοι, ε, βρίσκεται σε αναταραχή αυτή την εποχή. Κάνουν απεργία πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί ακριβώς κινδυνεύει η ίδια τους η ύπαρξη, η ίδια ελευθεροτυπία. Τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι στους οποίους αναφέρομαι εργάζονται για εξευτελιστικά μικρά ποσά, είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, προσπαθούν να ανέβουν, προσπαθούν να βρουν μια πιο καλοπληρωμένη δουλειά. Έχει όμως ε, αποδειχθεί αδύνατον. Πλέον γίνεσαι δημοσιογράφος μόνο αν ε, ο μπαμπά και η μαμά σου πληρώσουν τις σπουδέ, σου πληρώσουν μαθητεία για κάποια χρόνια, αμυστή σε κάποια εφημερίδα. Και αυτές οι μαθητείες ε, συνεχίζονται Νομίζω πως οι πιο επιτυχημένοι εκδοτικοί οίκοι προσπαθούν να επεκταθούν ακόμα περισσότερο, προσπαθούν να πάρουν το κομμάτι της πίτας που ανήκει στους ε, μικρότερους και το κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει να τους ε, προστατεύσει. Όπως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, που κάποιος δηλαδή υπογράφει ότι δίνει όλα του τα δικαιώματα στον ε, εκδότη, διαφορετικά δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βέβαια κάποιες προτάσεις σχετικά με τη διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Χρειάζεται να γίνουν όμως πολλά περισσότερα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους ε, δημοσιογράφους, να προστατεύσουμε όσους ασχολούνται με την βιομηχανία του θεάματος έτσι ώστε να ε, συνεχίσει να υφίσταται ο κλάδος. Χρειάζεται λοιπόν το Κοινοβούλιο να προστατεύσει αυτόν τον κλάδο του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χόλτερνες. Κύριε Ντόνταντς έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Είναι σωστές κυρία Φαρέν αυτά που είπατε. Πάντα μπορεί κανείς να αγοράσει όλα τα περιεχόμενα μιας εφημερίδες, οποιοδήποτε και να είναι, σε οποιοδήποτε τομέα, όπως λέτε. Τώρα, η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον, μπορείτε σε μία έντυπη έκδοση να έχετε διαφορετική δυνατότητα. Και όπως είπατε κι εσείς, είναι εύκολο να πωλήσει κανείς κάτι στον αναλογικό κόσμο σε κάποιον, αλλά στον ψηφιακό είναι δύσκολο ένα άρθρο να το πωλήσετε εσεί, να του βάλετε δηλαδή τη δική σας, ε, ε, το δικό σας τίτλο, δική σας υπογραφή και να το πωλήσετε σε κάποιον. Είναι δύσκολο να έχετε τέτοιου είδου και να ζητήσετε πληρωμή. Και βεβαίω αυτό σημαίνει ότι οι νέε εφημερίδε έχουν λιγότερε σελίδε από ό,τι αυτές του παρελθόντες. Εμείς αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε, διότι έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις και πρέπει να πω και στον τομέα το δικό μας βεβαίως γίνονται και στον τομέα αυτό μεγάλες επενδύσεις και οι επαφές μας και με τις διάφορες επιχείρησεις έχουν σχέση με αυτό το δεύτερο ερώτημά σας τώρα κυρία Φερχάινεν αφορούσε τα δικαιώματα των εκδοτών Στη Γερμανία το 2013 ο Γερμανός νομοθέτης μερίμνησε για αυτά τα θέματα, τα δικαιώματα δηλαδή των εκδοτών. Ίσως θα θυμάστε κάποια στοιχεία. Μετά από την εισαγωγή αυτού του νόμου ζητήσαμε στην VGD ε, Media να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας. Μετά αντέδρασε η Google και όλοι οι εκδότες της VG Media ε, ότι θα πρέπει να ζητούν κάποια δικαιώματα, διαφορετικά η Google θα ε, τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν οι υπεύθυνοι των ε, διαφημίσεων για να μην ε, υπάρχει ε, μείωση των εσόδων του να προσαρμοστούν. Είπανε λοιπόν νομοθέτες ότι δεν ε, έσπασε τους κανόνες του καρτέλ η Google και βεβαίως η λύση που βρέθηκε δεν ικανοποίησε τους πάντες αλλά εμείς σταματήσαμε τις συμβάσεις με το VG Media για να στείλουμε μήνυμα στη Βρυξέλλες. Δηλαδή να πούμε, αν θέλετε, όντως, να σταματήσετε αυτή την πρακτική, θα πρέπει να μην επαναλάβετε τις, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίσαμε εξαιτίας της γερμανικής νομοθεσίας κατά την απόψή μας, λαμβάνοντας υπόψη τι έγινε στην Γερμανία, πιστεύουμε ότι η νομοθεσία της που προτείνει τώρα η Κομισιόν θα είναι καλύτερη από τη δική μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, λέει ο τρίτος Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση της ε, κυρίας Κώστα για την ε, ε, ευθύνη των εκδοτών και το πώς μοιραζόμαστε ε, το ρίσκο και τις κοινέ πλατφόρμες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, είναι διαφορετικό από... και να το εξετάζουμε χωριστά από την σχετική οδηγία που ασχολείται με αυτό το θέμα. Επίσης, το σχόλιο για τον κανόνα του 20% εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς κάναμε τη δική μας ανάλυση και είμαστε σίγουροι ότι ευελιξία που επιτρέφει αυτό το 20% θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις δαπάνες διαφήμισης για τον τομέα των εντύπων. Θα θέλαμε το θέμα αυτό να παραμείνει έτσι όπως είναι στην ε, σχετική οδηγία ΒΕΟΜΕΣ. Τώρα, πώς μπορεί κανείς ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, να τα κάνει να είναι πιο σοβαρά στην εκπαίδευση, να εκπαιδεύσει περισσότερο. Κάποια. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει σχέση μεταξύ δημοσιογράφων, ε, σχολείων, μαθητών για να τους μάθουν να διαβάζουν, να μελετούν καλύτερα, να μάθουν ίδια να γράφουν άθρα, να μεταλλεύονται τι ικανότητες που έχουν για να βοηθούν το δικαίωμα. Προσχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά το copyright, σας είπε ο συνάδελφος Ντούντουνς πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσατε να είμαστε εδώ, να ακούσετε τις ιδέες μας και να σας πούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και πώς αναπτύσσεται ο τομέας μας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ήταν πάρα πολλές σαφείς οι παρουσιάσεις σας. Μας είπατε τι ακριβώς θα θέλατε, πώς θα θέλατε να ε, εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι ενεχόμενοι και άλλοι οι οποίοι φορεί που έχουν άλλα συμφέροντα στον τομέα. Εν πάση ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και κάνατε τις ε, παρεμβάσεις σας και μας εξηγήσατε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε την ημερησία μας διάταξη Λοιπόν, συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Έχουμε δύο ακόμα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Πριν περάσουμε λοιπόν το θέμα της απαλλαγής, θα ήθελα απλώ να σας πω ότι ο συνάδελφος Τζαμπάσκης δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί γιατί δεν είναι καλά σήμερα, έχει γρήπη και δεν μπορεί να μιλήσει, ε, κλείσει τη φωνή του. Και επειδή δεν υπάρχει συνάδελφος από το ECR που θα μπορούσε να τον αντικατασταήσει, θα ήθελα να σα ζητήσω να συμφωνήσουμε το εξή. Την επόμενη εβδομάδα να λάβουμε την εκθεσή του, ε, να υπάρχει χρόνος ε, βέβαια, μα πιέζει λίγο η ημερήσια διάταξη και μόλι το μάθαμε ότι δεν θα έρθει θα είναι λίγο πιο ε, στενή η προθεσμία για τις τροπολογίες. Δύο μέρες μετά την παρουσίαση της επόμενης συνεδρίασης. Δεν έχουμε άλλη λύση γιατί δεν υπάρχει κανείς από το ECR και δεν είναι εδώ και ο συνάδελφος. Μόλις τώρα μάθαμε ότι δεν θα μπορέσει να έρθει, επομένως η μόνη λύση είναι να το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Αν συμφωνείτε να περάσουμε τώρα στην απαλλαγή, την ε, γνωμοδότησή μου για την απαλλαγή για το 2015. Γνωρίζετε ότι αυτή τη φορά είμαι αρμόδια για τη γνωμοδότηση. Είδατε την πρόταση που υπέβαλα, το σχέδιο γνωμοδότησης. Το 2015 ήταν η δεύτερη χρονιά της εφαρμογής του νέου πολιτούς δημοσιονομικού προγράμματος και είναι προφανές από το 2015 ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων, κυρίως η Ευρώπη για τους πολίτες και η Δημιουργική Ευρώπη και γι' αυτό και επεσήμανα ότι πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί η πρικοδότηση εκεί. Για το Erasmus Συν Γνωρίζετε ότι το 2015 είχε σταματήσει στην Ελλάδα το έργο που αφορούσε την νεολαία, αλλά μετά ευτυχώς ε, έγινε μία ανάκληση της αναστολής ε, το 2016. Επισήμανε επίσης πολύ σημαντική δουλειά της ΑΤΣΕΑ για το τι ακριβώς έγινε ώστε να είναι να μπορούμε να τα παρουσιάσουμε και διαδικτυακά κάποια προγράμματα. Ε, για κάποιους βέβαια υπάρχει ακόμα πολλή γραφειοκρατία και υπάρχουν ε, αρκετές δυσκολίες και δεν μπορούμε να έχουμε και τα γραφεία να συμμετέχουν στην βελτίωση των συστημάτων ε, και της στρατηγικής. Όσον αφορά τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουν ζητήσει και οι ενδιαφερόμενοι και είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε γιατί το 2015 είχαμε αρκετέ επιφυλάξει όσον αφορά τους τρόπου πληρωμής. Το πρόγραμμα για το, η μόνιμη χρηματοδότηση του 2013 και το πρόγραμμα για την νεολαία ε, είχαν θέματα με τις ε, χρηματοδοτήσεις και υπήρξε αίτημα και πρόταση να γίνεται καταποκοπήν πληρωμή των ε, παραδεκτών πληρωμών και όχι μόνο τμηματικές πληρωμές, ώστε να διευκολύνουμε λίγο και τους δικαιούχους. Αυτό το προτείνουμε να τεθεί σε εφαρμογή και εφαρμόστηκε το 2015 και υπάρχει και ένα πρόβλημα που αφορά τα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελών, τα οποία έχουν ε, υπερπληθώρα μαθητών και θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ε, υπάρχει και ένα πέμπτο πλέον ευρωπαϊκό σχολείο από το ε, ε, σχολικό έτος 2019-2020. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο περιθώριο, αλλά βέβαια ε, θα ε, υποβάλω και κάποιες ερωτήσεις, έχω κάποιες επιφυλάξεις εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους σκιώδεις ή τις διάφορες πολιτικές ομάδες, ε, διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό για το 2015. Η Πέτρα Καμερέδε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια για την γνωμοδότησή σου. Πιστεύω πως η απαλλαγή είναι μια τυπική διαδικασία, όμως μπορούμε να κάνουμε και κάποιες προτάσεις, κάποιες μικροτροποποιήσεις. Να πω εδώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μας επέστησε στην προσωπή, την προσοχή στον αριθμό των ε, απορριφθέντων ετοιμάτων από τους πολίτες, για, για τους πολίτες. Πιστεύω πως εδώ φαίνονται τα προβλήματα που έχουμε. Σίγουρα είναι απόλυτα σωστά αυτά που είπες και να μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό ε, πως αυξήθηκαν τα κονδύλια για, τα το Erasmus Plus. Αυτό έγινε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις ε, στον τριμερή διάλογο. Καταφέραμε όμως παρά τις ε, δυσκολίες να έχουμε αυτή την αύξηση. Δεν φτάνουν όμως, δεν φτάνουν τα χρήματα. Αναγκαζόμαστε να απορρίψουμε πάρα πολύ ωραίες ιδέες, πάρα πολύ καλά έργα, ακριβώς γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Και θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα κονδύλια που έχει λάβει παραπάνω το Erasmus να μην διατεθούν σε κάτι περίεργα προγράμματα και έργα τύπου Interrail κτλ. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά πρέπει να ε, κάνει και εκείνη τη δουλειά της, ε, να δει τι μπορεί να αλλάξει στο Erasmus έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε κονδύλια. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι στο Erasmus Plus να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους Ευρωπαίους. Ναι, ναι, συμφωνώ ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να το υπενθυμίσουμε αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα ε, στην πραγματικότητα αυτά τα λεφτά τα οποία προβλέπονται δεν υπάρχουν. Ε, υπάρχουν μόνο 50 εκατομμύρια. Μόνο 50 είναι εκατομμύρια ε, στην πραγματικότητα για το 2017. Δεν είναι όσα προβλέπονται. Συνολικά, ναι, ναι. ναι συνολικά, ναι, όχι τα επιπλέον. Εντάξει, εντάξει. Ε, θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε στους στόχους του Εράσμους και να μην χρησιμοποιηθεί το Εράσμους ως ταμείο για να κάνουμε άλλα πράγματα. Ε, αν ε, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια. Ο κύριος Στρογέσκη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, κυρία Κώστα, και να πω ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε μόνο το 1 τρίτο ε, που ε, ασχολείται με προϋπολογισμό. Έχουμε την Κομισιόν, έχουμε το Συμβούλιο. Αυτό όμως ε, το 30% θεωρώ πως είναι λίγο. Αποφασίζουμε για ποσοστώσεις οι οποίες είναι πολύ μικρές. Βλέπουμε πως έχουν αρχίσει υποχωρήσεις από το σχέδιο Juncker στο οποίο σχέδιο Γιούνκερ βλέπουμε μια δραστική μείωση των κονδυλίων για τον πολιτισμό και μια γενικότερη απροθυμία. Όμως, βλέπουμε ότι τώρα εμφανίστηκε και ο πολιτισμός ε, με τη μορφή της ε, δημιουργικής βιομηχανίας και πως υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα διατεθούν εκεί. Αυτό όμω είναι μόνο δεν υπάρχει ακόμα κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Δεύτερον, υπήρξαν και προτάσεις να κλείσουμε το πρόγραμμα Erasmus Plus, να σταματήσει. Και καταφέραμε να το σώσουμε, καταφέραμε αυτή τη στιγμή να μην απειλείται η ύπαρξή του, ε, έχει βελτιωθεί και η ρευστότητα του προγράμματος. Σίγουρα δεν είναι πολλά τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας, όμως νομίζω πως ε, δεδομένης της ε, κατάστασης δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου τα όσα έχουμε καταφέρει να, καταφέρει να κερδίσουμε. Είχαμε πολλές διαφωνίες με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι όσα και αν ζητάμε στο τέλος αυτά που θα πάρουμε είναι ελάχιστα. Τώρα, αν θα ονομάσουμε το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Ευρώπη για πολίτε, Erasmus Plus, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να απαιτήσουμε περισσότερα κονδύλια για πιλωτικά προγράμματα. Ας δούμε τι, θα γίνει μάλλον το 2017. Του χρόνου λοιπόν είναι βελτιωμένα τα πράγματα από την κατάσταση την οποία περιγράφει η παρούσα γνωμοδότηση. Όμως δεν πρέπει να θεωρούμε πως είναι ικανοποιητικό αυτό, διότι τα κονδύλια παραμένουν πολύ χαμηλά για όλο τον προπολογισμό. Μάλιστα θα τολμούσα να πω ότι απλά έγινε μία αναπροσαρμογή ε, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Πρέπει να προσέξουμε εδώ την διαφορά στάσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις κρατών στην Ένωση, οι οποίες ε, είναι και τα φιλόδοξες ε, ως προς τον ε, πολιτισμό και τα σχέδια που έχουν. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προγράμματα. Μέχρι το 2015 όμως μόνο οι μισές κυβερνήσεις είχαν αναγνωρίσει ότι ο πολιτισμός χρειάζεται κονδύλια. Η Ελλάδα ήταν ένα άσχημο παράδειγμα. Όμως υπάρχουν και άλλα τέτοια άσχημα παραδείγματα, τα οποία ε, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Α, κατά τα άλλα δεν έχω κάτι να πω. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλες παρεμβάσεις. Ε, να σταχυολογήσω κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Εγώ σας είπα ότι θα πρέπει να προτείνω και κάποιες τροπολογίες. Είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας βέβαια. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι από το 2015 ε, δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα στην Ευρωπα... Ε, δημιουργική Ευρώπη το νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο ήρθε αργότερα. Να σας το υπενθυμίσω γιατί θα χρειαστεί και αυτό φυσικά. Θεωρώ ότι το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μπορούμε να το συνδέσουμε σε αυτό, στις επενδύσεις για τον πολιτισμό, γιατί ε, καταφέραμε και κάτι με την ε, Δημιουργική Ευρώπη και Μία δέσμευση που είχε ε, κάνει ο Επίτροπο Έτιγκερ με την πλατφόρμα για τη δημιουργική Ευρώπη να μπορούσαμε και μέσω του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων να συμπεριλάβουμε και τα κονδύλια για το νέο ε, χρηματοδοτικό μέσο για τη δημιουργική Ευρώπη. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά τόσο το Εράσμους, αλλά τον τίτλο 3, τη Δημιουργική Ευρώπη και την Ευρώπη των Πελιτών, διότι και φέτος αποφασίσαμε να επιμείνουμε να αυξηθεί το ανώτατο όριο του ε, τίτλου αυτού, διότι τώρα έχει τη μετανάστευση, την ηθαγένεια. Τελικά δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες. Ε, ε, έγιναν κάποιες κινήσεις, αλλά ελάχιστα ήταν. Χρειαζόμαστε περισσότερα λοιπόν. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις τροπολογίες, η προθεσμία είναι για το... Δεκεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου συγγνώμη στις 11 και στις 24 Ιανουαρίου Ψηφίζουμε τώρα. Επειδή όπως σας είπα ο συνάδελφος Τζαμπάσκι δεν μπορεί να παρευρεθεί, ε, όπως είπαμε αναβάλλεται το θέμα του για την επόμενη συνεδρίαση. Ε, δεν θα υπάρχει μεγάλη προθεσμία για τροπολογίες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, 3 με 6.30. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας βράδυ.